Um, Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Είχα ένα πρόβλημα με τον ενελκυστήρα και άλλοι θα έχουν προβλήματα με τα σανσέρ λοιπόν. Οπότε θα γεμίσουμε σιγά σιγά την αίθουσα. Σήμερα το πρωί έχουμε την Επίτροπο Κρούζ η οποία ήρθε για να μας ενημερώσει για θέματα ανταγωνισμού θα κάνουμε το εξής. Η Επίτροπος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Μετά από αυτό θα υποβληθούν ερωτήσεις. Και ανάλογα με το πόσοι θα ενδιαφερθούν ή θα απαντηθούν μία-μία οι ερωτήσεις ή σε ομάδες. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Αν το πρόβλημα των ελκυστήρων είναι το μόνο σημερινό πρόβλημα, καλά θα ήταν. Είναι χαρά που είμαι μαζί σας. Και ενδιαφέρομαι για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας διαγραφήσω τα τεκτενόμενα. Ξεκινώ συγχαίροντάς σας για την ε, επανεκλογή σας, για την εκλογή σας. Είναι καλή παράδοση που αναλαμβάνουν θέσεις οι γυναίκες. Είμαστε σε καλή θέση και σας εύχομαι πολύ τύχη. Με καλέσατε για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας για το 2008. Πριν όμως ξεκινήσω, θα προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την παρούσα κρίση. Είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει. και παρέλαβα κάποιες τις παρατηρήσεις σας. Θυμάμαι που είπατε ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον κίνδυνο και να τον εξαφανίσουμε. Συμφωνώ, συμφωνώ. 100% αλήθεια είναι. Χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας, μεγαλύτερη αυτοπιθαρχία. Είναι λογικό, είναι κομμάτι της λύσης. Αυτοπιθαρχία αυτή αυτή δεν μπορεί να μας απαλλάξει και να μας, από τα προβλήματα και να μας οδηγήσει στην επίτευξη στο στόχο μας που είναι η νέα αγορά. Είναι η κορονίδα των προσπαθειών μας. Αυτή η κρίση εν γέννη αντιμετωπίστηκε όχι πολύ άσχημα εν συγκρίση με τη μεγάλη ύφεση του παρελθόντος και τις μεγάλες απειλές του προστατευτισμού. Είχε κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιστάθηκε στον προστατευτισμό και προστατεύσαμε την ενιαία αγορά μέσω του ανταγωνισμού, του ελεύθερου. Ήταν μεγάλη όμως η χρηματοπιστωτική κρίση και διαπιστώθηκε ότι διαμορφώνεται μια άλλη τάση. Και εδώ αναφέρομαι στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκόλυνε κάποιες προσπάθειες. Λοιπόν, επεκράτησε μια σύγχυση μετά την κατάρρευση των Lehman Brothers Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζε και τα κράτη-μέλη με έναν κάπως καινούριο τρόπο ούτω ώστε να επικρατήσει η νομική ασφάλεια για να εξευρεθούν λύσεις και να επιβληθεί κάποια σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιδράσει στην κρίση συνδυάζοντας κοινοτικές πολιτικές ήταν κρισίμου σημασίας. Χρησιμοποίησαμε τις εμπειρίες μας από νομισματική και οικονομική πολιτική και τις χρηματοστικές αγορές για να διαμορφώσουμε μέσω πολιτικής ανταγωνισμού την απάντησή μας. Και μας βοήθησαν συνάδελφοι για την εφαρμογή, μάλλον βοηθήσαν συναδέλφους να διαμορφώσουν πολιτικές μέσω του ανταγωνισμού. Και αυτό αποδεικνύει πόσο καλό είναι να έχουμε κάτω από μία αιγίδα όλες αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπω όλα τα συστήματα και το δικό μας μπορεί να βελτιωθεί. Μετά όμως από χρόνια προσπαθειών βελτιώσεω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύστημά μας είναι αποτελεσματικό τουλάχιστον. Πολλοί το θεωρούν ως το καλύτερο ε, σύστημα, αλλά είμαστε μετριοπαθείς. οι έλεγχοι κρατικών ενισχύσεων τόνισαν αυτή την εικόνα και από την αρχή της εντολής μου προσπάθησα να διαμορφώσω αυτή την πολιτική κρατικής ενίσχυσης και ευτυχώς μπορώ να πω ότι κινηθήκαμε εγκαίρως. Και τότε υπήρξε μεγάλη υποστήριξη για την στρατηγική και πολιτική μας τη μακροπρόθεσμη για ανάπτυξη και απασχόληση. Μέχρι ότου ξεκινήσει η κρίση, τα κράτη-μέλη πράγματι δαπανούσαν λιγότερα στις ενισχύσεις αλλά είχαν ε, περισσότερα κέρδη, διότι μέσω οριζοντίων μέτρων, ανάπτυξη, καινοτομία κλπ. είχαν στοχεύσει αυτή την ενίσχυση για να βοηθήσουν τις βιομηχανίες που είχαν προβλήματα και τις τομείς που είχαν προβλήματα. Και χαίρομαι που από την αρχή της θητείας μου ακολουθήσαν αυτή την προσέγγιση. Διότι όταν ήρθε η κρίση έστειλε τους οικονομολόγους στο μηδέν, στην αφετηρία και ήταν σημαντικό να βρεθεί μια ειδική απάντηση. Τέσσερα χρόνια μεταρρυθμίσεων, κυρία Πρόεδρε, έδωσαν τη δυνατότητα να βρούμε καλύτερη απάντηση, να αντιδράσουμε καλύτερα και είδαμε ότι πολλές ενισχύσεις δόθηκαν σε ξεχωριστές τράπεζες. Μπορεί η ενίσχυση να πήγε σε τράπεζες, όμως για να επιτευχθεί οριζόντιος στόχος, η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αυτός ο οριζόντιος στόχος ήταν, αποτέλεσε και ένα από τα μεγαλύτερα βήματα πρόοδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Κινούμεθα μέσα σε κρίση. Χρειαζόταν ευελιξία και ταχύτητα. Πετύχαμε το στόχο μας χωρίς να υπονομεύουμε την αρχή των ισότιμων συνθήκων ανταγωνισμού. Ούτε ζητήσαμε επιταγή εν λευκό από τους φορολογούμενους. Ήταν μεγάλα τα προβλήματα του περασμένου έτου και είναι επίτευγμα το ότι η ενιαία αγορά ε, παρέμεινε ακέραιη. Είναι γεγονός αυτό και χρωστάμε πολλά, πολλές ευχαριστίες στο, ενίο, στο μοναδικό μας σύστημα ανταγωνισμού. Αν έπρεπε να κατατήσω έναν κατάλογο που θα περίχει αυτό που μας βοήθησε σε αυτή τη χειρότερη φάση της κρίσης, θα έλεγα ότι υπάρχουν ε, οι εξουσίε για άμεση επιβολή, το σωστό θεσμικό πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμότη μέσω συνεχών μεταρρυθμίσεων, λειτουργών δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού και κύρος, καλή φήμη αν θέλετε και προθυμία να τίθενται τα σωστά ερωτήματα και δέσμευση για συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη, για συνεπή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Πιστεύω όμως ότι ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση και δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τις θεμελιώδεις, τα θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού μας μοντέλου. Όπως σίγουρα θα παρατηρήσατε σε πρώτερα σχόλιά μου, ένα βασικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στην ετήσια έκθεση είναι ότι χρειάζεται συνδυασμό σταθερών αρχών με ευέλικτες διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι που μας βοηθά να περάσουμε την κρίση. Και με μεγάλη χαρά σημειώνω ότι και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μας βοήθησε πάρα πολύ στις προσπάθειες. Έχουμε προσωπικό που ασχολείται με τις συγχωνεύσεις και τις πολιτικές κρατικών ενισχύσεων στον ίδιο χώρο, στον ίδιο τομέα και αυτό είναι λογικό. Στον τομέα των τραπεζών. Συλλέγουμε τις γνώσεις, ομαδοποιούμε τις γνώσεις και αυτό συνέβαλε σημαντικά σε ποιοτική και ταχύ απάντηση και η δυνατότητα να εστιαζόμεθα επί συγκεκριμένου θέματος ή τομέα θα μας βοηθήσει εξίσου για να βγούμε από την κρίση. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφέρω ένα-δύο μέσα πολιτικής. Μετά από προτάσεις που έγιναν στην έκθεση των Αθηνών, η ετήσια έκθεση του 2008 συμμετέχει περισσότερες λεπτομέρειες και οι πληροφορίε είναι φιλικότερε για τον χρήστη, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μα το είχατε θίξει πέρσι. Δηλαδή, μέτρα αναδιάθρωση, διάσωση, βελτίωση όσον αφορά την καταπολέμηση της κρίσεω. Χρειάζεται ξεκάθαρη επικοινωνία. Αυτό σημειώθηκε. Το παρατηρήσαμε. Το περιλάβαμε και σε έγγραφα προσανατολισμού που μας οδήγησαν σε προσπάθειες καταπολεμήσης της κρίσης, κατευθυντήριες γραμμές για τα, τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών, αναδιάθρωση τραπεζικού τομέα, αυτά που συμφωνήσαμε Φεβρουάριο και Ιούλιο και πρέπει να προχωρήσουμε με τα εν λόγω σχέδια. Οι προσανατολισμοί υπάρχουν και πρέπει τώρα να δράσουμε. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 έχει παραταθεί ο προσανατολισμό μα για την κρατική ενέσχυση, η διαδιάσωση και αναδιάθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εκδώσαμε νέε κατευθυντήριε γραμμέ και οδικού χάρτε ούτω ώστε να διοχετεύονται σωστά τα δημόσια χρήματα προ τα προγράμματα που μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά από όλου του πολίτε. Επίση, προβλέπεται κατάρτιση, ενίσχυση για κατάρτιση σε άτομα με αναπηρία και που είναι σε δυσκερή θέση. Και υπήρχε ε, τότε πολιτική ε, πίεση να αρθούν οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Πάντα ήμουν σαφής. Η οικονομική ανάπτυξη σημαντική για τον ανταγωνισμό. Και σε μια κρίση πρέπει πάντα να το εξηγούμε ότι είναι λογικότερο μάλλον κατά τη διάρκεια κρίσεως να δούμε ότι ο ανταγωνισμό επιτρέπει καλύτερη κατανομή των πόρων, προστατεύει του καταναλωτέ και προστατεύει και του φορολογούμενου. Και εξασφαλίζει ο ανταγωνισμό δυνατότητε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τονώνει και την καινοτομία. Και θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να πούμε ότι ήταν ειδική περίπτωση ο χρηματοστικό τομέα. Ουσιαστικέ παρεμβάσει στον χρηματοστικό τομέα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ω δικαιολογία για μαζικές κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άλλους τομείς. Και καμιά φορά το δοκιμάζουν αυτό, αλλά εγώ ε, είμαι άκρος αρνητική. Δεν είναι διότι μας νοιάζουν περισσότερο οι τραπεζίτες από τους εργαζομένους άλλους τομείς, αντιθέτως θα έλεγα, αλλά διότι το χρηματοστατικό ε, ο τομέας είναι το κυκλοφοριακό του συστήματός μας. και ωφελεί την οικονομία. Σωστή εφαρμογή πολιτικής ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσης σε όλους του τομείς είναι βασικό στοιχείο για ταχύ ανάκτηση των οικονομιών μας χωρίς να σπαταλάμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Και είμαι σίγουρη ότι κι εσείς ε, δέχεστε πιέσεις από τους συμπολίτες σας, τους ψηφοφόρους που σας ρωτούν τι κάνετε με τα χρήματά μας τα χρήματα των φόρων μας. Τι υποστηρίζετε, τι δεν υποστηρίζετε. Όσον αφορά την ανάκαμψη, θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία που θεωρώ λογικά. Πιστεύω ότι απέχουμε πολύ από τη λήξη της κρίσης. Εκείνοι που λένε ότι περάσαμε την κρίση, ότι βγήκαμε, νομίζω ότι ονειρεύονται θα πρέπει να δεχτούμε τα οικονομικά, την οικονομική κατάσταση επί σειρά ετών και κυρίως όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Και συμφωνώ με τον ΟΣΑ, διότι η σημερινή κρίση και οι σχετικές πολιτικές δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη, ούτε την ενία αγορά να την υπονομεύσουν. Σας διαβεβαιώ ότι το πλαίσιο του Τάμπερε για τις κρατικές ενισχύσεις εξυπηρέτει σημαντικό σκοπό και εξακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να κρατήσει αυτό το πλαίσιο του Τάμπερ, τα προσωρινά μέτρα έχει του Τάμπερ, ζητώ συγγνώμη. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι θα κάνουμε τα δέοντα χρησιμοποιώντα τα προσωρινά μέτρα. Πολλές πρωτοβουλίες ανελήφθησαν όσον αφορά τον έλεγχο συγχωνεύσεων και το θέμα των trust και τους κανόνες antitrust Προβλέπονται δικασίες διευθετήσεων, κατευθυντήρες γραμμές για την επιβολή των διατάξεων όσον αφορά ε, δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεων και τις ε, κοινοποίησεις όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που αφορούν τις συγχωνεύσεις. Τώρα χρησιμοποιούμε τις έρευνες του τομέα με νέες έρευνες. Βλέπουμε τι γίνεται με τον γεράσκοντα πληθυσμό με τις απειλές όπως είναι η γρήπη των χείρων. Πρέπει να βελτιωθεί του σχετικού τομέα. Και είναι σημαντικό, κυρία Πρόεδρε, να σημειώσουμε ότι η τομιακή έρευνα αποδίδει καρπούς επί σειρά ετών. Όπως στον τομέα της ενέργειας. Αυτοί παρακολούθησαν τα τεκτενόμενα στον τομέα της ενέργειας, θα το γνωρίζουν αυτό. Λοιπόν, περιμένετε καινούρια μαντάτα τους επόμενους μήνες. Η έκθεση του 2008 συμπεριλαμβάνει εστιασμένα κεφάλαια για τα καρτέλ και για τους καταναλωτές. Και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχετε καθορίσει για την καταπολέμηση των καρτέλ, τα πρόσφατα στατικά στοιχεία τι μας δείχνουν. 34 επιχειρήσεις 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 περιπτώσεις καρτέλ το 2008 τομέα μπανανών, ό,τι θέλετε, διάφοροι τομείς καλύπτονται. Οκτώ επιχειρήσεις, 1,24 δις σε δύο υποθέσεις του 2009. Δεν έχει τελειώσει όμως η χρονιά, όπως ξέρετε. Και προσπαθούμε να δούμε τι βλάβες δημιουργούν τα καρτέλ. Και είναι ενδιαφέρον και καμιά φορά ο κόσμος θεωρεί τι έχετε βρει, ποια είναι τα πορίσματά σας αυτή είναι η καλύτερη σας μέρα, η καλύτερη μου μέρα θα είναι ότι θα έχουμε επιβάλει μηδενικά πρόστιμα. Αυτά ήταν πρόστιμα που σας προανέφερα. Θέλουμε να έχουμε μηδενικά πρόστιμα. Αλλά απέχουμε πολύ από το τέρμα. Δεν υπάρχουν αγγελούδια στον πλανήτη. Λοιπόν, προσπαθούμε να προσμετρήσουμε τη βλάβη που προξενούν τα καρτέλ. Πρέπει να καταλάβουν όμως και οι πολίτες καλύτερα τι γίνεται μπορούν να γίνουν περισσότερα. Αυτή είναι η αρχή. Οι, Ευρω... οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασαν 18 καρτέλ που υπόκειται σε αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στο 2005 και 2007. Χρησιμοποίησαμε υποθέσεις πολύ συντηρητικέ. 10% υπέρβαση όσον αφορά τις βλάβες, υπερεκτίμηση. 7,6 δις ήταν για τα 18 καρτέλ. Με αυτή την υπερεκτίμηση του 10% κάμψη υπολογισμού μα. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στου καταναλωτέ. Πρέπει να του πούμε. Θέλετε να συνεχίσει αυτό. Ή θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγάλος ο λογαριασμός για τους καταναλωτές. Και σίγουρα τα πραγματικά στοιχεία είναι πολύ ψηλότερα. Βάσει έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι για κάθε καρτέλ που ανακαλύπτεται ίσως να μην έχουν δημιουργηθεί πέντε καρτέλ ή να μην έχουν εγκαταλειφθεί πέντε καρτέλ. Και αν αυτό το εφαρμόσουμε, το πόρισμα, σε όλη την εσωτερική αγορά, βλέπουμε ότι η δουλειά μας για τα καρτέλ γλιτώνει δεκάδες εκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων. Τι επικρίσεις ακούσαμε όσον αφορά τις διαδικασίες και τα πορίσματα. Για τα καρτέλ και όλοι οι άλλοι παραβάτες βλάπτουν όλους. Τα καρτέλ βλάπτουν τους πάντες. Χρειάζονται αποτρεπτικά μέτρα για να μειωθούν οι βλάβες αυτές στο μέλλον. Κάποιοι μου λένε ότι είναι υπέρ των ε, καταναλωτών αυτά τα υψηλά πρόστιμα και κατά των επιχειρήσεων. Δεν συμφωνώ με αυτό. Και οι εταιρείε υποφέρουν από το μεγαλύτερο κόστος εάν οι προμήθευτές τους δημιουργήσουν καρτέλ. Αποτρεπτικά μέτρα είναι υπέρ και όλων των νομίμων επιχειρήσεων. Και οι περισσότερες επιχειρήσεις, η τεράστια πλειοψηφία αυτών, είναι νόμιμες. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό, να το ξεκαθαρίσω. Και κάποια πρόστιμα είναι μεγάλα, αναμφισβήτητα. Αλλά πάντα σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών των εταιριών, τα προϊόντα που παράχθηκαν, τις υπηρεσίες που παρεδόθηκαν και το μέγεθος της παράβασης και τη διάρκεια αυτής. Ποτέ δεν ξεπερνάμε το 10% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, τα πρόστιμα. Και για κάθε πέντε πρόστιμα καρτέλ έχουμε λιγότερο από 5, επιβάλλεται πρόστιμο λιγότερο από 5% του ετησίου κύκλου των ε, επιχειρήσεων. Είναι αποτελεσματικό ε, αποτεπτικό μέσο οι, ποινέ αυτά τα πρόστιμα, αλλά ε, μα, γλιτώνουμε ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων χρόνο. Έχοντας αυτά υπόψη, σας παρακαλώ να εξετάσετε τις λεπτομέρειες και μην διαβάζετε τι επικεφαλίδε όσον αφορά αυτό το θέμα. Μπείτε στι λεπτομέρειε, για καταλάβετε. Εν κατακλείδη, θέλουμε να είναι ισότιμες οι συνθήκε ανταγωνισμού και να αυξηθεί ε, το θετικό κλίμα για τον καταναλωτή. Αλλά έχουμε και το έργο μας έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα. Δείχνει ότι στεναρή ρύθμιση είναι εφικτή και εκείνοι που κλέβουν το σύστημα αποδεικνύεται ότι θα τιμωρηθούν. Αυτό δείχνουμε. Και αυτό είναι ένα ούκα σήμαντον μήνυμα. Όχι μόνο για αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική, αλλά και για τους λαούς, για τους πάντες στην Ευρώπη. Και εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πέτυχε όλα αυτά για, για ένα κόστος κάτω από 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Βλέποντας τις συνέπειες μου στην αγορά και συγκρίνοντας με τα δισεκατομμύρια των ζημιών που γλιτώσαμε από τα καρτέλ και αυτούς που καταχρώνται την αγορά, βλέπουμε ότι η ανταγωνιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματικά είναι, έχει αξία, αποδίδει. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. We've taken to ε, χειροκροτούμε τους ομιλητές για τα σχόλιά τους και εμεί ευχαριστούμε επίσης για το ρόλο σας ε, στην ε, οικονομική κρίση διότι ξέρουμε ότι δεν ήταν εύκολο ο κανείς ε, να κρατήσει μια σταθερή γραμμή σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις και φαντάζομαι ότι αυτό θα το θίξουν και άλλοι διότι όπως είπατε ε, υπήρχαν διάφορα βασικά ε, βασικές φάσεις οι οποίες ε, μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Εσείς καλύπτετε τον καταναλωτή και αναφερθήκατε εις τις ζημίες που προκάλεσε η Λευκή Βίβλος και επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ε, τι έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τωρινή της ε, εντολή και την προηγούμενη φορά επίσης μας είχατε πει ότι θα εμπλέξετε το Κοινοβούλιο όσο μπορείτε περισσότερο ή στην ε, εργασία σας πράγμα το οποίο συνέδραμε το Κοινοβούλιο πριν τις εκλογές οπότε νομίζω ότι ε, εφόσον αυτή, αυτό το πρώτο θέμα ήταν βασικό για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεώρησα ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι λαμβάνουν υπόψη ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλη την ομάδα των ε, οικονομικών ε, υποθέσεων ε, αισθάνομαι ότι έχω μία υποχρέωση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα πρέπει να σας ενημερώνω βαθμιαία, θα πρέπει να ενημερώνω τα μέλη της Επιτροπής και πλέον αυτού θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό που ανεφέρθη στην έκθεσή σας ήταν ένα σαφές μήνυμα το οποίο μελετήσαμε και όντως τώρα μπορούμε να πούμε ότι μας βοήθησε στον τρόπο που σκεπτόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει μελετήσει την, ε, το ψήφισμά σας για τη Λευκή Βίβλο. Δεν θέλω όμως να επαναλαμβάνω αυτά που έχω ήδη πει ε, και πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο πρεσβεύετε. Άρα ε, το, <coughs> στα θέματά μας δεν πρέπει να υπάρχει ομαδική προσφυγή, class action. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε ε, τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε θα σας ε, συμβουλευτούμε προτού εφαρμόσουμε ό,τι οι αποφάσεις λαμβάνονται και ε, θα θα πρέπει να πω ότι κατά την προηγούμενη πενταετία έχουμε λύσει και τα ευρωπαϊκά προβλήματα αλλά και ε, τα θέματα που εξετάζονται συλλογικά στη Λευκή Βίβλο. Θα είμαι λοιπόν σε στενή επαφή μαζί σας και ελπίζω ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένετε προλή για την αντίδρασή μας ε, θα κάνουμε τώρα ερωτήσεις σε ομάδες των τριών και ε, η πρώτη ερώτηση είναι από έναν αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς την ίδια ερώτηση ήθελα να θέσω στην κυρία Επίτροπε. Η κρίση κάνει ότι τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα και αυτή είναι η είδηση η χθεσινή και η προχθεσινή είδηση είναι ήδη παρελθόν και σε χθεσινή είδηση με, σε σχέση με μια επιστολή από την Ισπανική κυβέρνηση όσον αφορά τον Επιτροπό με κάποια σημεία. Δηλαδή η διάσωση open θα πρέπει να γίνει με κριτήρια εμπορικά και οικονομικά αποκλειστικά. Και δεύτερον, η Μάγνα, εκείνος ο οποίος αγόρασε την Opel, πρέπει να κάνει την καλύτερη χρήση των μέσων όχι προχθές αλλά κάποιες μέρες πιο πριν είχαμε την είδηση ότι οι G20 αποφάσισαν λέει προανήγγυλαν ότι η έξοδος από την κρίση πρέπει να είναι συντονισμένη δράση και όχι κάθε χώρα ξεχωριστά με τα δικά της μέσα. Η ερώτηση είναι, θεωρεί η Επίτροπος ε, ότι θα πρέπει να κρίνεται για την συνεκτικότητα ή όχι των επιχορηγήσεων που έχουν υποσχεθεί οι Γερμανοί για τη διάσωση της Όπελ που πρέπει να γίνει αποκλειστικά με κριτήρια ανταγωνισμού. Η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η διάσωση της Όπερ πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια αποκλειστικά βιομηχανικά ή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετες ε, σκέψεις, ε, κάποια πρόσθετα στοιχεία. Και επιπλέον θα μπορούσε να διασυνδεθεί η χορήγηση αυτών των επιδοτήσεων με τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε κάποια βιομηχανία, σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ευχαριστώ. Uh, Κυρία Βότμαν Κόλ, παρακαλώ, επόμενη. Yeah, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα, αν επιτρέπετε, να εκφράσω την εκτίμησή μου κύριε Επίτροπε για το γεγονός ότι εσείς πάντα προσέρχεστε εδώ στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και είσαστε πρόθυμοι για διάλογο μαζί μας. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω για την οδηγία, για την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των τραπεζών. Πώς κρίνετε ε, περιπτώσεις πριν από τον Ιούλιο Είχατε πει ότι αναπερίπτωση θέλετε να αποφασίσετε τι θα γίνεται. Δεν θεωρείτε όμως ότι για αυτές τις δράσεις υποστήριξης ε, θα πρέπει πραγματικά επίσης να υπάρχουν κάποια αυστηρά κριτήρια αν τώρα γίνεται η προσπάθεια η ING να περάσει μέσα σε ε, κάποια κριτήρια υπό την προϋπόθεση του Ιουλίου 2009, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα ισχύσουν. Εσείς νομίζω εξετάζετε την έδρα των τραπεζών ποια είναι. Θα πρέπει όμως επαρκώς ε, να, δούμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε διεθνώς ένα ε, level playing field, ένα ισότιμο πεδίο δραστηριοτήτων. Υπάρχουν ε, θυγατρικέ ή έδρε στις ΙΦΑ. Δεν θεωρείτε ότι όταν πρόκειται κάποια τμήματα επιχειρήσεων να απολυθούν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται θα πρέπει να ανακτηθούν τα χρήματα αυτή της τεράστια πελώριας δράση. Έχω την εντύπωση ότι παράλληλα με τους στόχους σας έχετε υπόψη σας και ένα άνοιγμα της αγοράς όπου η αγορά ήδη σήμερα είναι μία από τις πιο ανοιχτές θα έλεγα παγκόσμια λέγεται λαμβάνοντας υπόψη ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ε, να λάβετε αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος παρακαλώ τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε η θητεία σας θα λήξει σύντομα. Έχετε την ετήσια έκθεση που υποβάλλεται, δείχνετε τι έχετε κάνει. Είναι σημαντική η πολιτική για τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Υπό τι κατηγορίε των ε, κρατικών επιδοτήσεων, τη απαγόρευση ε, των καρτέλ και των ελέγχων συγχωνεύσεων έχετε πάρα πολλέ ε, εξουσίε και αρμοδιότητε. Αυτό το οποίο παρατήρησα σε αυτή την πενταετή σχεδόν θητεία σας και θέλω να το αναφέρω αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει. Στον τομέα της ενέργειας, ενεργειακό τομέα, έχει παρέμβει στην τρέχουσα νομοθεσία, στην εξελίξει νομοθεσία. Αυτό το θεωρώ μια επέμβαση στι αρμοδιότητε τη αρχής για τα ενεργειακά θέματα. Δεύτερον, οι κατευθυντήριες γραμμές, ε, οι διατάξει ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής βασίζονται σε μια ανεδαφική βάση στον κανονισμό 17 του 1965 του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος συναπόφασης ή εμπλοκής της Ευρωβουλής ε, και συναπόφασης. Πρέπει να αναθεωρηθεί λοιπόν αυτό το πλαίσιο αυτής της νομικής βάσης. Και πέρα από αυτό, τομεακά πρέπει όλες τις περιπτώσεις να εξετάσετε. Ακόμα και αν ένα κράτος μέλος ε, έχει κάποιες διαμαρτυρίες ή αιτήματα όσον αφορά την Όπελ, εντάξει, βαίνει, καλό αυτό, αλλά να χρησιμοποιήσετε αυτά ως ε, έτοιμα για να ανατραπεί ένας ολόκληρος τομέας είναι εκπληκτικό, με εκπλήσει αυτό. Τώρα λέτε πρέπει ο τομέας των φαρμακοβιομηχανιών να, να εξεταστεί. Ε, αυτό είναι το τελευταίο θα έλεγα, ε, η τελευταία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Υπάρχουν προβλήματα να βρεθούν όλο και νέα τεκμήρια ή ε, δικαιολογίε. Θα ήθελα να μα πείτε τι συμβαίνει. Θέλουμε να συναποφασίζουμε ω Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για κατευθυντήριε γραμμέ και θέματα αρχών. Ευχαριστώ. Επίτροπε, θα θέλατε να απαντήσετε στις πρώτες αυτές ερωτήσεις. Η Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη και ο Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ σωστά ανέφερε πιο πριν ότι οι επιστολές πραγματικά αποστέλλονται από τα κράτη-μέλη και όχι μόνο από την Ισπανική κυβέρνηση εντάξει αλλά και από άλλες έχουμε αριθμού, κρατημέλη που επικεντρώνονται στα ίδια θέματα και ακόμα και αν ήταν και μόνο η Ισπανική κυβέρνηση τότε πάλι θα υπαρκούσε πρέπει να πούμε για να λάβουμε εμείς υπόψη ότι πρέπει να είμαστε σαφέστατοι για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και να κρυθούν να αξιολογηθούν. Θεωρούμε, θε, θυμάμαι πάντα τις συζητήσεις στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο όταν συζητούσαμε το τι διακυβεύεται ακριβώς. Και θα έλεγα όταν κάνουμε λόγο για ένα προσωρινό πλαίσιο το οποίο θα ισχύει και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις το είπα ότι υπήρχε νόημα για την ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου για εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες ακριβώς που ε, παρόδο επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από την οικονομική κρίση και αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ώστε να δοθεί μια διέξοδο στα κράτη-μέλη ακολουθώντας πάντα τις συστάσεις ε, της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης καταλήξαμε στην έγκριση αυτού του προσωρινού πλαισίου στήριξης. Εφαρμόζοντας, εκτελώντας αυτό το προσωρινό πλαίσιο στήριξης, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν οποιονδήποτε τομέα με ευνοϊκούς όρους. εξού και την αυτοκινητοβιομηχανία. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ο κύριος στόχος μας φυσικά είναι να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Μια πάρα πολύ σημαντική βιομηχανία αυτή για την Ευρώπη, χωρί αμφιβολία. Πάρα πολλέ θέσει απασχόληση, ε, πάρα πολλά οικονομικά προτερήματα απορρέουν από την ύπαρξή τη εδώ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι είναι μια βιομηχανία με υπερπλεονάζον δυναμικό, υπερβολικό δυναμικό. Το προσωρινό λοιπόν αυτό πλαίσιο στήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν μια εταιρεία η οποία έχει πληγεί δεν είχε ε, προηγούμενα πριν από την κρίση εμπλακεί σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια στήριξη. Και έτσι υιοθετήσαμε τη γραμμή ότι η διαχωριστική γραμμή του Ιουλίου 2008 ήταν η διαχωριστική γραμμή τελικά. Για την επιστροφή και στους κανονικούς κανόνες όσον αφορά ανάκτηση και αναδιάρθρωση και αυτό το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ισότιμο πεδίο δράση. Πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, α το πω έτσι, οι στρεβλέ δράσει. Και πρέπει να καταλήξουμε και απαντώντα σε αυτέ τι ερωτήσει και από πλευρά Κοινοβουλίου και από αυτήν την ερώτηση που διατυπώσατε εσεί, τοποθετούμε και λέω ότι κάτι τέτοιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο να συμβαίνει, με κάθε σαφήνεια το λέω, όταν πραγματικά δεν είναι πολιτικά τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη Ούτε γεωγραφικές λοιπόν, ούτε άλλες ε, σκέψεις ή στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αφορούν τα κριτήρια ανταγωνισμού φυσικά τα οποία αναφέρατε. Τώρα, γεγονότα, συμβάντα, στοιχεία ακλόνητα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία επιλέγουμε και στα οποία βασιζόμαστε. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τη γερμανική, γερμανική κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σε κάποια ερωτήματά μας σε σχέση με τις ε, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την περίπτωση Όπελ της General Motors. Λαμβάνοντας πάλι επίσης υπόψη ότι κάνουμε λόγο εδώ για θέσεις απασχόλησης, αλλά όχι μόνο θέσεις απασχόλησης σε ένα κράτος μέλος, είναι ευρωπαϊκή αυτή η προοπτική, αυτή η πρόκληση, ας το πω έτσι, να βρούμε μια λύση. Στο τέλος, θα, πρέπει να είναι μια βιώσιμη βιομηχανία αυτή και μια βιομηχανία στραμμένη προς το μέλλον με δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν δέχομαι μια βραχυπρόθεσμη, κοντόθωρη προσέγγιση που θα διασφάλιζε μόνο κάποιες θέσεις απασχόλησης βραχυπρόθεσμα. Πρέπει μακροπρόθεσμα να το δούμε, να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνε που έχουμε υπομειστεί. Τούτων λεχθέντων, στη συνέχεια, δεν υπάρχει λευκή εν λευκό επιταγή που υπογράφεται με κανένα τρόπο. Δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, μια εντάχει απόφαση που λαμβάνεται και βιαστικά να πούμε να δώσουμε το εντάξει για να προχωρήσει κάτι. Κάνοντας λόγο για την ING τώρα. Εδώ πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο, ας το αποκαλέσω έτσι. Το... Πάρα πολλά συμβαίνουν σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και διαφορετικά θέματα. Πρώτον, ένεση κεφαλαίου. 10 δις ευρώ θα αποδεχθεί, θα δοθούν στην ING. Το εγκρίναμε αυτό τον προηγούμενο Νοέμβριο. Το 2009 πήρε κρατικές επιχορηγήσεις η ING και πάλι σε σχέση με μια μελέτη impact assets μεταφέροντας ε, και όσον αφορά τα θέματα πετρελαίου στην, ε, στο Ολλανδικό κράτος ε, και σε ύψος 21 δις. Περί τίνος πρόκειται τώρα εδώ συνολικά. Αποδεχθήκαμε εμείς προσωρινά τις τα μέτρα αυτά όσον αφορά το impact το 2009 και μετά ανοίξαμε το burden sharing. Η αξιολόγηση, η αποτίμηση του μέτρου αυτού δημιούργησε κάποιες ε, αμφιβολίες και η προσωρινή αδειοδότηση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου παρατάθηκε και ταυτόχρονα παρατάθηκε η σε βάθος εξέταση των πραγμάτων αυτού του χαρτοφυλακίου. Περί τίνος πρόκειται εδώ, τι διακυβεύεται εδώ. Έχουμε έντονες ισχυρές αμφιβολίες και το αποκαλώ, το λέω διπλωματικά, αν η αξιολόγηση αυτού του χαρτοφυλακίου μπορεί να θεωρηθεί συνετή και σόφρον. Και όλα αυτά συνδέονται φυσικά με τη δική μας ευθύνη δική μας ευθύνη. Κάνουμε λόγο εδώ για κρατικές επιχορηγήσεις, έτσι, για ένα ισότιμο δίκαιο πεδίο δραστηριοποίησης. Και βλέποντας εδώ τα όσα τεκταίνονται και είναι ενδιαφέροντα εδώ και ένα χρόνο, υπάρχουν δόξα τω Θεώ υγιείς τράπεζες και υγιείς τράπεζες από αυτό το κράτος μέλος που με τις, μπορούμε να πούμε ότι με τις εξετάσεις ε, που κάνουμε μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει βαίνει καλός ο, ο τομέας, ανακάμπτει, εξηγένεται, είναι προς όφελος όλων, αλλά πρώτον πρέπει να υπάρχει ένα ίσο και δίκαιο πεδίο δραστηριοποίησης για όλους και πρέπει σε σχέση με τους ανταγωνιστές, με τα κονδύλια φορολογουμένων, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις ε, και χρέη. Και αυτό είναι η κατευθυντήρια γραμμή για την αναδιάρθρωση των τραπεζών και την προσαρμογή. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στο τέλος τέλος ότι υπάρχουν ε, επιπτώσεις στο τέλος. Είναι ίσως κάπως δυσάρεστο για κάποιες τράπεζες αυτό όμως τι να κάνουμε. Το θέμα της προσαρμογής και της υποβολής μετά ενός λογαριασμού που πρέπει να πληρωθεί και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα να διασφαλίσουμε μια ειφορία για το μέλλον και να διασφαλιστεί αυτή η βιωσιμότητα για τον τραπεζικό τομέα στο μέλλον και λέγοντας είμαστε υπέρ τη ανοιχτή αγορά στην Ευρώπη, τέλεια, συμφωνώ με αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε όμω και σίγουρα θα χρειαστούμε ισχυρού παίκτε που θα δρουν σε αυτό το πεδίο, μια και κάνουμε λόγο για παγκοσμιοποιημένε αγορέ. Η αξιολόγηση, η αποτίμηση λοιπόν του χαρτοφυλακίου είναι ένα θέμα και πρέπει να λάβουμε σίγουρα υπόψη ότι υπάρχουν επιπτώσεις για τη χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων και πρέπει αυτά να εμπλέκονται όλα σε αυτά τα οποία εμείς εγκρίνουμε εν τέλει. Και όσο το δυνατόν γίνουν ταχύτερα αυτά και διευθετηθούν, τόσο το καλύτερο. Θα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και των περιπτώσεων που εξετάζουμε. Τώρα, ο κύριος Λάγκεν έκανε λόγο για τα ενεργειακά, στο πω εσύ, θέματα. Πραγματικά, εμείς είχαμε προηγούμενα στο παρελθόν συζητήσεις σχετικά και ξεκινήσαμε με, τον, με την ε, εξέταση διακρύβωση του τι γίνεται στον ενεργειακό τομέα. Και είδαμε ότι εδώ θα πρέπει να δούμε τα θέματα των κρατικών ε, ε, επιδοτήσεων. Και συνδυασμένα, όχι μόνο για τον σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει νόημα αυτό και για τους συναδέφους επιτρόπους και για τον Άντρες ε, Πίμπαλξ και για το Σταύρο Δήμα για θέματα περιβάλλοντος να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις πτυχές ε, που μας εμπλέκουν στον ενεργειακό τομέα. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις εξέτασης λοιπόν είχαμε κάποιες περιπτώσεις ώστε στο τέλος να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα η αγορά και να διασφαλίζεται αυτό και οι ε, καταναλωτές να υποφελούνται από τα ωφέλη που απορρέουν. Τώρα κάνοντας λόγο για την Όπερ, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ στην απάντηση προς τον Αντιπρόεδρο προηγούμενα που έδωσα, πραγματικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό Εκεί πρέπει να δούμε τα θέματα υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού και όχι με πολιτικά κριτήρια τα οποία μπορούν να επηρεάζουν μια λήψη απόφασης. Και μια άλλη παρατήρηση θα ήθελα επίσης να προσθέσω. Νομίζω πραγματικά σε σχέση με τα θέματα ανταγωνισμού θα πρέπει να ε, υπάρχει δυνατότητα να ληφθεί με ιδιαίτερο τρόπο από πλευράς της διαχείρισης η, ο ανταγωνισμός υπόψη. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο δεν ακούστηκε. Η προσωπική μου πείρα κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ως Επιτρόπου είναι ότι πραγματικά δεν είναι μόνο ένα θέμα του να είμαστε συνεπείς ε, και συνεκτικοί όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, τα δημοσιονομικά, αλλά και σε άλλους τομείς το ίδιο. Και είμαι βεβαία ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εσείς προτείνετε για περαιτέρω εξετάσεις ε, περιπτώσεων στο μέλλον θα είναι μια πρόκληση πραγματικά να δούμε ποιος τομέας πρέπει να εξεταστεί. Και για τα φαρμακευτικά εμείς θεωρούμε πραγματικά, βρήκαμε πραγματικά ότι κάτι γινόταν και σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον τομέα που δεν τέριαζε στην δική μας προσέγγιση για θέματα ανταγωνισμού και γι' αυτό το εξετάσαμε. Και όταν εσείς ε, κάνατε ένα σχόλιο σε σχέση με το κόστος για την υγεία και τον προϋπολογισμό για τα θέματα υγείας και σε σχέση με τους πολίτες της Ευρώπης λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι για παράδειγμα ο αυθόδης πυρετός των χείρων που επηρέασε αυτή την υπόθεση παραμένουμε πιστοί σε αυτά και αυτή τη στιγμή κάνουμε λόγο για μια μεγάλη α το πω εσύ υπόθεση και έχω υπόψη ότι κάνοντας λόγο για τέτοια πράγματα έχουμε κόστος το οποίο δεν μπορούμε να, να μας επιβαρύνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διευθέτηση, εξυγίανση αυτού του τομέα και να βρεθεί ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να προαγάγουμε τον τομέα αυτό όπως και σε, άλλα, σε άλλους τομείς ε, υιοθετώντα πρακτικές που από πλευρά των εταιριών ε, θα εξοικονομήσουν κόστος. Και είμαι βεβαία ότι θα είμαστε σε επαφή και θα σας ενημερώνουμε για τα τεκτενόμενα σε σχέση με αυτόν τον τομέα επίσης. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομάδα των τριών, Μπόλμαν, Πρεσάδο και μετά ο κύριος Γκοζές και μετά πάλι Επίτροπος. Ο κύριος Μπούλμαν λοιπόν παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή πάντα υποστήριζε μια ισχυρή πολιτική για τον ανταγωνισμό. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Ακριβώ στην κρίση που προαναφέρατε πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρά ενιαία και συνεκτικά με ολοκληρωμένε προσεγγίσεις πολιτική και θα πρέπει να κατέβει από τα θεωρία και να δει τα θέματα για την λύση τη Όπελ. Όπελ λοιπόν. Στα πρώτα χρόνια της θητείας σας, 10.000 θέσεις απασχόλησης αποκλειστικά από την ε, General Motors στη Γερμανία χάθηκαν. Τώρα διακυβεύονται 50.000 θέσει απασχόληση στι θηγατρικέ τη General Motors και δημιουργεί μια γέφυρα η γερμανική κυβέρνηση. Γιατί δεν λέτε εσεί από την βιομηχανική πολιτική εντάξει να διατηρήσουμε, καλό είναι, τι βιομηχανίε αυτέ στην Ευρώπη, να υπάρχει μια δυνατότητα νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη. Φυσικά πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχέ τη πολιτική του ανταγωνισμού. Αλλά θα ήθελα να μα πείτε ποιο είναι το πρόγραμμά σα, πότε θα ολοκληρώσετε αυτό τον έλεγχο, τι εξετάσει για να μην πάνε στραβά τα πράγματα υπό τη βιομηχανική πολιτική. Χρειαζόμαστε γοργά μια σωστή προσέγγιση. Πρέπει όμω ένα μέρο των πολιτικών λύσεων βιομηχανικά να τι δώσετε, γιατί αλλιώ θα χάσουμε το παιχνίδι. Μετά, όσον αφορά το επόμενο θέμα, εσεί για την Πολωνία δίνετε μια ε, επιχορήγηση 54 εκατομμυρίων στην Πολωνία σε μια περιφέρεια. Ταυτόχρονα από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση έχουμε το κλείσιμο ή την απόλυση 2.000 εργαζομένων στην Ιρλανδία με 14 εκατομμύρια ή παραπάνω από 14 εκατομμύρια και η Ντέλ αγοράζει για κάποια δισεκατομμύρια δολάρια ε, εταιρείε. Ποια είναι αυτή η συνεκτική ολοκληρωμένη πολιτική. Δεν υπάρχει. Μπορούμε να προσθέσουμε και παραδείγματα της Νόκια και άλλων επιχειρήσεων. Πού δράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βιομηχανική πολιτική και την περιφερειακή πολιτική ολοκληρωμένα και με ένα συνεκτικό τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν βλάβε και στρεβλά αποτελέσματα αριστερά ή δεξιά. Αυτό θα ήθελα να μα πείτε. Είμαστε υπέρ μια ισχυρή πολιτική για τον ανταγωνισμό. Ε, είμαστε είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και να μην κάνουμε λάθη και να μας παραπλανούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που συνεργαζόμενοι κάναμε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Χρηματοοικονομική κρίση. Δεύτερον, για τα, ε, ε, ε, τον ιδιωτικό τομέα και τον γαλακτοκομικό τομέα τρίτο. Είδαμε εδώ ότι εδώ η σταθερότητα και ο ανταγωνισμός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την χρηματοοικονομική κρίση. Ο ανταγωνισμός έχει ρόλο να διαδραματίσει, αλλά έχουμε μεγάλη πορεία να καλύψουμε ακόμα. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Χρειάζεται κάποιο διάστημα, αλλά πρέπει να δούμε τις στρατηγικές εξόδου. Αναφέρομαι σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια έχουμε και τα θέματα των εγγυήσεων, πρέπει να δούμε τα θέματα των επενδύσεων, να δούμε τα θέματα ε, περιορισμών και να, δούμε, να, να αποκλείσουμε να επαναληφθούν τέτοιου είδου ε, μη αηφόρα προγράμματα ή τέτοιου είδου εγχειρήματα που δεν θα είναι αηφόρα. Αναφερόμενο ε, στι ιδιωτικέ επιχειρήσει και τα στην, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που ομόφωνα εγκρίθηκε, εξετάστηκε ότι θα πρέπει να συναποφασίζει το Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει η διαβούλευση. Εδώ πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα και πρόκειται για δικαιώματα των καταναλωτών. Και για όλου του λόγου και για την νομική ασφάλεια επίση και νομική βεβαιότητα θεωρούμε ότι υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάζονται αυτά, υπό τη συναπόφαση. Για το γαλακτοκομικό τομέα ζήσαμε μια πολύ σημαντική κρίση με κατάρρευση των τιμών. Είμαστε όμω μάρτυρε ότι σε σχέση με τι τιμέ που, που δίνονται στου παραγωγού δεν υπάρχει αναλογία στι τιμέ ε, για του παραγωγού και στι τιμέ καταναλωτών ετών. Ε, έπεσαν 50 ε, και παραπάνω τις 100 οι τιμές ε, για τους παραγωγούς και λιγότερο οι τιμές για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει λοιπόν αναλογία και έτσι αυτό είναι προς ζημία των παραγωγών. Και σίγουρα και ζημιώνονται και οι καταναλωτές. Πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχει επικέντρωση παραγωγής και δεσπόζων ρόλων, πριτανεύων ρόλος κάποιων. Δεν πρέπει να παρέμβεται στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να κυνηγήσουμε αυτούς που είναι ζαβολιάριδες αλλά πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ και διστάζω όταν μας λέτε ότι τελικά ε, θεωρητικά το δόγμα του ανταγωνισμού πρέπει να είναι προς όφερος του καταναλωτή αλλά πρέπει να υποχωρήσει ε, σε σχέση με την εργασία και την απασχόληση γιατί αν δεν υπάρχει απασχόληση δεν υπάρχει καταναλωτής οπότε μου κάνουν ε, ε, έκπληξη τα, τα σχόλιά σας στην ε, Νέα Υόρκη αλλά ήταν το γραπτό κείμενο δεν ξέρω αν τα ίδια είπατε και προφορικά θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε δύο θέματα καταρχήν στην επιλεκτική στην επιλεκτική εφαρμογή για τις ε, εταιρείες πολυτελείας και δεύτερον όσον αφορά την οδηγία για τις ε, υπερβολές της αγοράς. Δηλαδή πρόκειται ε, να υποβληθεί ένα σχέδιο ενώ υπάρχει μία συζήτηση με τους ενδιαφερομένους για τις ομαδικές προσφυγές διότι δεν ε, πρέπει να επιβαρύνει κανείς τις εταιρείες με θέματα τα οποία είναι εις βάρος της ή στην περιοχή τους. Η Επίτροπος, θέλετε να απαντήσετε και να προσπαθήσετε να είστε πιο σύντομοι γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα ε, και ξεκινώ από το τέλος δεν θα υπάρξει προσέγγιση όπως στις Ηνωμένε Πολιτείες διότι ε, ε δεν ε, δεν μπορώ να προχωρήσω. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ε, εφαρμογή της ομαδικής προσφυγής και δεύτερον ότι ε, το πρόβλημά μας ε, θα πρέπει να επιληθεί βάσει του σεβασμού των κανόνων ανταγωνισμού διαφορετικά θα το πληρώσουμε ακριβά διότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική Ευρώπη αλλά και μια Ευρώπη με υγιή βιομηχανία και βιομηχανία βιώσιμη βιομηχανία και αυτό είναι μια από τις προκλήσεις της κλίσεως. Ε, θα πρέπει να υποφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας για να δούμε πόσο μπορείτε να αποκαταστήσετε την δυνατότητα της βιομηχανίας να επιβιώσει και η αυτοκινητοβιομηχανία δεν πρέπει να συνεχίσει με την υπερβολική προσφορά και ε, να μην ανταποκρίνεται εις τους κανόνες της ζητήσεως και της προσφοράς. Επίσης Υπάρχει το παράδειγμα της Dell θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα αλλά με την ε, ε, ε, περιφερειακή ενίσχυση και με άλλες ενισχύσεις θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν αυτά τα οποία θέλουν να κινήσουν στην οικονομία τους αλλά στην περίπτωση της Dell και αυτό μου το έχουν πει οι ίδιοι υπεύθυνοι της Δέλ που θα πρέπει να προσήγησαν και εσάς ε, σκόπευαν ούτως ή άλλως να φύγουν από την Ιρλανδία οπότε το θέμα δεν είναι αν έχουν περισσότερη χρηματοδίτηση ή όχι ήθελα να κινηθούν εκτός Ευρώπης και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο είμαι ευγνώμων διότι έχουμε τη δυνατότητα της περιφερειακής ενισχύσεως που επέτρεψε στην Πολωνία να υποδεχθεί αυτές τις βιομηχανικές δραστηριότητες ε, το έχουμε συζητήσει και προηγουμένως κυρία Πρόεδρε διότι μια απόφαση του επιχειρηματικού κόσμου δεν είναι καταρχήν βασισμένη στο πόσο θα ενισχυθούν από κρατικέ ενισχύσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ε, η ποιότητα της εργασίας σε ένα κράτος μέλος, η υποδομή το φορολογικό σύστημα και ούτω καθεξής. Οπότε διαπιστώσαμε από την έκθεση η οποία καταρτίστηκε κατά την Γερμανική Προεδρία οπότε ε, ζήτησε η Γερμανία από μια εταιρεία συμβούλου να προβούν στην έρευνα και διαπιστώσαμε ότι η κρατική ενίσχυση είναι η 13η νομίζω προτεραιότητα. Άρα δεν είναι ένα θέμα του ότι θα έφυγαν για κάπου αλλού, θα έφευγαν με την Λανδία ούτως ή άλλως. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι δεν δραστηριοποιούμαστε μόνο στι αναδιαρθρώσεις αλλά επίσης και ε, ε, για να ε, λύσουμε άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε τώρα στη δεύτερη φάση στην αναδιάρθρωση αλλά θα υπάρξει και μία τρίτη βαθμίδα και καλό θα είναι να εφαρμοστεί σύντομα όταν μιλάμε για την αναδιάρθρωση της αγοράς πρέπει να ξέρουμε ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί την κορονίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο τα 27 κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν Οπότε όταν μιλάμε ε, για τις ε, ε, ομαδικές προσφυγές θα σας ενημερώσω. Ξέρω τι θέλετε, αλλά δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Ελπίζουμε όμως να τα καταφέρουμε. Επίσης, ένας άλλο θέμα το οποίο ε, συζητήθηκε ε, Ξέρουμε βέβαια ότι οι γαλακτοπαραγωγοί υποφέρουν αυτή τη στιγμή και το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ποιος παίρνει την αφρόκρεμα διότι χωρίς, ε, χωρίς καμία αμφιβολία θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ε, να ε, ικανοποιήσουμε το ε, θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τα γαλακτοκομικά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που πολλές φορές έχουν περισσότερα θέματα που διακυδεύονται παρά εμείς και επίσης υπάρχει ένας κατάλογος μέτρων για να ενισχύσουμε τις ε, γαλακτοβιομηχανίες και εμείς θα πρέπει να προβούμε σε μελέτες τομεακές και να συνεχίσουμε τις έρευνές μας για την κατάσταση της αγοράς αυτής. Η, Επιτροπή, πολιτική ανταγωνισμού θέτει σε πρώτη θέση ε, τους καταναλωτές, τους καταναλωτές που θα καταναλώνουν, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας και γι' αυτό εδώ θέλουμε να έχουμε βιώσιμες ε, βιομηχανικές δραστηριότητες διότι μόνο όταν ε, η απασχόληση δεν εξαρτάται από τις κρατικές ενισχύσεις μπορούμε να την ε, εγγυηθούμε ώστε να υπάρξει απασχόληση και μετά από μία δύσκολη περίοδο. Τώρα όσο αναφορά τις πωλήσει μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ε, στην τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα έχουμε ένα συνέδριο για τους ε, ε, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και θα ασχοληθούμε και με τις πωλήσει της μουσικής μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα εξετάσουμε διότι βλέπουμε ότι υπάρχει 30% ε, κύκλος εργασιών στις πωλήσει αυτές και ε, θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις ε, είναι, ξεκινάμε τη Σόφη Έντβελτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, δεν πρόκειται ε, μόνο για την παρουσία σας στην ε, Επιτροπή αυτή που σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά όμως καταρχήν να κάνω μια γενική, ένα γενικό σχόλιο, διότι πολλές φορές έχετε την εντύπωση ότι ορισμένοι θεωρούν ότι η πολιτική ανταγωνισμού οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασία. αλλά αυτό οφείλεται μάλλον όταν η βιομηχανία δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα σύγχρονα κρατούντα και χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Δεν είναι δηλαδή ε, κάτι το οποίο σχετικά με τις κρατικές ε, ενισχύσεις πρέπει να εξεταστεί μόνο από τη σκοπιά της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να έχω απαντήσεις και μία πιο λεπτομερή ανάλυση για το πόση ε, κρατική ενίσχυση μπορεί να δοθεί και πόσο σημαντική είναι. Διότι αν δείτε την έκθεση ανταγωνισμού που καταρτίστηκε πέρυσι, πολλά στοιχεία αναφέρονται, αλλά ε, ιδίω πρέπει να εξετάσουμε βάσει ε, ποιων στοιχείων έχετε απορρίψει ορισμένες αιτήσει, διότι σε κρατικές ενισχύσεις θα αποδοθούν στην αυτοκινητοβιομηχανία και πολλοί μπορεί να πούν ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα, τους πόρους αυτούς για να εξασφαλίσουμε ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω και αυτό είναι μία από τις ερωτήσεις που απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να δούμε ε, εάν χρησιμοποιούν κρατικές ενισχύσεις για αυτήν την ε, ριζική αλλαγή προς το καλύτερο περιβαλλοντολογικά πράσινα ή όχι. Δεν είμαι βέβαιη. Μιλήσατε επίσης για τις πωλήσει μέσω του διαδικτύου και επαναλαμβάνω αυτό που είχε πει ε, η έκθεση Εύα για τον ανταγωνισμό πέρυσι ότι ζητήσαμε να υπάρχει ε, ε, είχαμε εξετάσει το θέμα των διαφημίσεων διότι πολλές εταιρείες έχουν μια πολύ στεναρή ε, θέση από αυτού του θέματος. Καταρχήν θα ήθελα να διασφαλίσω και πάλι ότι υπάρχει υποστήριξη διότι οι, ε, γερμανικοί, γερμανοί καταναλωτές υποφέρουν από τα ολιγοπόλια και είναι καλό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μέτρα σε αυτό το τομέα διότι δεν μπόρεσε να το πράξει η, γερμανική πολιτεία μέχρι στιγμής. Ε, έχω όμως και μία άλλη ερώτηση σχετικά με το σχόλιο που κάνατε στην ε, νοτιοανατολική, ε, ε, νοτιογερμανική βιομηχανία προκαιρού όπου είπατε ότι οι συνθήκες είναι πεπαλαιωμένες και δεν ανταποκρίνουν το ρόλο που πρέπει να παίζει η Γερμανία σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω τι εννοείται και αυτό συνάδει με το γεγονός ότι πρέπει να προωθήσετε τον ανταγωνισμό και όχι να τον μειώσετε διότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι καλύτερο να έχουν δυνατότητα ε, να προσφύγουν σε χρηματοδότηση από, διάφορα, από διάφορες μορφές τραπεζών και όχι από λίγες μόνος. Επίσης ε, ε, οι μεγάλες τράπεζες όντως χρηματοδοτήθηκαν με μεγάλα ποσά ενώ οι συνεταιριστικές τράπεζες χρειάστηκαν να βρουν αλλού χρηματοδότηση. Επίσης όσον αφορά την αποταμίευση και τα αποταμιευτικά ιδρύματα εποφελήθηκαν από τα μέτρα σας και τέλος όσον αφορά τα φορολογικά. Θα ήθελα να ξέρω το εξής. Υπάρχουν πολλά μέτρα άνισου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ο κώδικας συμπεριφοράς για την φορολογία των επιχειρήσεων ε, δεν ακολουθεί και θα ήθελα να ξέρω αν πρόκειται να ε, χρησιμοποιήσετε την νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων και ε, πρόκειται να μπορέσουμε να έχουμε μία διέξοδο ανταγωνιστική από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και πάλι αναφέρομαι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχω και εγώ στείλει μια επιστολή στο γραφείο σας διότι υπάρχουν 5.000 ε, θέσεις που χάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο των οποίων 3.000 ε, είναι στην περιοχή μου, στο Λούτον. Χαίρομαι λοιπόν που λέτε ότι η ύφεση ε, δεν πρόκειται να δώσει ε, ε, την ελευθερία στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων εκ των οποίων επωφελούμασταν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν θεωρείτε ότι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή μου είναι αποτελεσματικές. Τι συγκεκριμένες πληροφορίες και ενέργειες αναλαμβάνετε αυτή τη στιγμή για να εξασφαλίσετε ότι οι κυβερνητικές ενισχύσεις όντως καταβάλλονται και όσον αφορά την αναδιάρθρωση η οποία δημιουργεί τεράστια βεβαιότητα όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τις οικογένειές τους οπότε θα ήθελα να θεωρήσετε το θέμα αυτό σαν πολύ επίγον και να μου δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα της ολοκληρώσεως της έρευνάς σας επ' αυτού του σημείου. Κύριε Επίτροπε, αν είσαστε έτοιμοι, σύμφωνα με την ε, Πράσινη Βίβλο, όσον αφορά ε, τις θέσεις εργασίας, τι είδος χρειάζεστε και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς η κρατική ενίσχυση. Ε, έχω έναν μακρύ ε, κατάλογο από τις εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αποδεκτές δεν είναι μόνο θέμα ε, αναδιαρθρώσεως του κεφαλαίου αλλά και άλλα μέτρα και ευχαρίστω θα σας ενημερώσω γιατί έχουμε ε, αποδεχθεί ε, το σύστημα των εγγυήσεων της αναδιαρθρώσεως του ενεργητικού μπορείτε να με ρωτήσετε δηλαδή τι δεν έχουμε αποδεχτεί αντί να με ρωτάτε τι έχουμε αποδεχτεί ε, θα μπορούσα να σας ενημερώσω αλλά είναι πάρα πολύ μακρύς ο κατάλογος για να τον παρουσιάσω τώρα όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία είναι ε, πολύ ενδιαφέρον διότι μιλάμε για μια υγιή ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη και να ξέρετε ότι πρέπει εκεί να προσθέσουμε και την πράσινη πρόκληση διότι είχαμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και ήταν μια δυνατότητα μέσω της οποίας μπορούσαμε να ενισχύσουμε ορισμένες προτάσεις αλλά τελικά ε, πιστεύουμε ότι θα είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε ε, περισσότερο και γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι οι εμπορικές ε, προϋποθέσεις τις οποίες λαμβάνεται υπόψη για εφαρμογή αυτού του είδους ε, κρατικών ενισχύσεων όπως στην περίπτωση Σόπελ παραδείγματος χάρη όσον αφορά τον τομέα της έρευνας ή την πρόταση εξετάσεως ενός τομέα που ανέφερε ένας συνάδελφός σας ε, για τις ε, διαφημίσεις στο διαδίκτυο ε, θα σας ενημερώσω τι έχουμε εντοπίσει αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον πλήρη κατάλογο. Ε, όσον αφορά τους Γερμανούς καταναλωτές, θέλω να σας πω ότι οι Γερμανοί καταναλωτές ε, μιλούσαν για ενέργεια η οποία ήταν πολύ ακριβή και μπορούσε να βελτιωθεί ε, διότι σε άλλα κράτη-μέλη ε, η κατάσταση ήταν διαφορετική και αυτό οφείλεται στο ότι οι μεγάλες εταιρείες εποφελόντουσαν τις δεσπόζουσες θέσεις τους. Αυτό είναι κάτι που καταφέραμε να σπάσουμε και ελπίζουμε ότι τώρα έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα και ότι τελικά ο, ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Όσον αφορά την δομή των τραπεζών στη Γερμανία και το σχόλιο που έκανα στη συνέντευξη που αναφέρατε, τελικά δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας τράπεζας, δεν με με το χολόγιο, αν ε, είναι κρατική τράπεζα ή ε, ιδιωτική και πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά ε, έχω άποψη αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ευθύνες που έχω αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν μιλάμε για ιδιωτικές τράπεζες, για συνεταιριστικές και για αποταμιευτικές ένα από τα μαθήματα τα οποία διδαχθήκαμε από την κρίση αυτή είναι ότι ο στόχος της τράπεζας και η πρόκληση για την τράπεζα είναι να μπορεί να δανείζει. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, ότι δηλαδή οι τράπεζες πλέον δεν ε, ε, καλύπτουν τις αρχικές τους ε, ευθύνες. Γι' αυτό και όταν μιλάτε ε, για τις επιχειρήσεις και για τους ιδιώτες ε, ο καθένας χρειάζεται να μπορεί να ε, βρει κοντά του μία τράπεζα η οποία μπορεί να τον δανείσει. Όταν μιλάμε όμως για τις Landesbanken ακόμη και τώρα σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα με τις Landesbanken. Δεν είναι ότι δεν βοηθήθηκαν από κρατικές ενισχύσεις αλλά δεν ήθελαν να επιβιώσουν και ο φορολογούμενος ε, ε, ίσως ε, δεν αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την κρατική ενίσχυση δεν θα επιβιώνανε, θα χρεοκοπούσαν άμεσα. Οπότε στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία και αλλού, αλλά είναι πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα στη Γερμανία, ε, οι συνεταιριστικές τράπεζες ουδέτερα πρέπει να επιβιώσουν αλλά σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού όχι χάρη σε κρατική ενίσχυση ε, θα πρέπει να βρουν μια διαφορετική διέξοδο ε, και ελέγχοντας την αγορά της, των λιανικών τραπεζιστικών δραστηριοτήτων διαπιστώσαμε από ε, τις ε, μελέτες μας ότι έπρεπε να μετρήσουμε ε, την δυνατότητα συνεργασίας και η διαδικασία της τραστ ε, κινητοποιείται όταν οι τράπεζες μεταξύ τους μοιράζονται τα μερίδια της αγοράς. Οπότε η κατάσταση των γερμανικών αποταμιευτικών τραπεζών ε, είναι συγκεκριμένη. Οι περισσότερες ε, είναι κρατικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και εσείς βέβαια ε, από ό,τι μου λέτε δεν συμφωνείτε ή τουλάχιστον αυτό μου δείχνετε με, την, ε, με τις κινήσεις σας αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι στη Γερμανία οι αποταμιευτικές τράπεζες έχουν μια ιδιάζουσα κατάσταση γιατί ελέγχονται ε, από το κράτος, από την τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, το οποίο για μένα είναι γεγονός και είναι συνειδιοκτήτες μαζί με τα κρατήδια της Γερμανίας που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και τώρα αναδιαρθρώνονται, είναι υποχρεωμένες να αναδιαρθρωθούν. Οπότε θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτές τις εξελίξεις όχι μόνο από πλευράς κρατικών ενισχύσεων αλλά και από πλευράς γενικότερης εμπιστοσύνης. Και τέλος, το, η τελευταία ερώτηση αναφερόταν σε φορολογικά θέματα. Ξέρετε ότι η συνθήκη δίνει τη δυνατότητα ή στην κοινότητα να μειώσει τις στρεβλώσεις ανταγωνισμού και ε, ορισμένα μέτρα φορολογίας των επιχειρήσεων όπως στο Βέλγιο παραδείγματος χάρη θεωρήθηκαν ως ε, ασύμβατες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάστηκε το κράτος μέλος που να τις καταργήσει. Όσον αφορά το, την περίπτωση του λούτων για την Όπελ στην Αγγλία. Σας είπα ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι εμπορική. Συμφωνώ. Επαναλαμβάνω αυτό που ήδη είπα. Τι κάνουμε λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία ιδέα μέσω αριθμών και γεγονότων για να καθορίσουμε ε, τις ενέργειές μας και όσο πιο γρήγορα θα τα έχουμε τόσο καλύτερα διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο πια αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν έχω τις απαντήσεις και εγώ όπως και εσείς αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται και έχουν θέσεις εργασίας εκεί και όχι μόνο μέσα στην Όπελ αλλά και οι διάφοροι προμηθευτές και γενικότερα, γενικότερα ολόκληρα χωριά τα οποία θα επηρεαστούν θα ζητούσαν και απαιτούν να υπάρχει μια γρήγορη επίλυση του θέματος. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη εκ προημίου. Πιθανότατα δεν θα μπορέσουν όλοι να παρέμβουν από αυτούς που το επιθυμούσαν. Η επόμενη ομάδα τριών, Ντανούτα Χούμπνερ, Σεκλούνερ και Χονγκόκ. Αυτή η κυρία Χούμπνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη εκτίμησή μου σε εσά Επίτροπε και στι υπηρεσίε σας για αυτό που κάνατε σε αυτή την περίοδο κρίσης. Δύο σύντομα αιτήματα έχω. Το πρώτο για τι τράπεζε, Γιατί ένα από του στόχου. Ε, της ε, οδηγίας της δράσης για τις τράπεζες ήταν να βοηθηθεί η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Χθε είχαμε μια συνάντηση με τον Ζαν Κλωτρίσε που είπε σαφώς και είπε ότι αναφέρεται ότι η οικονομική και νομισματική εξέλιξη είναι επιβραδυντική, επιβραδύνονται τα πράγματα ακόμα και σε σχέση με τις ε, ε, τους ισολογισμούς όσον αφορά τους ε, καταναλωτές, αυτό έχει επιπτώσεις. Η δική σας εκτίμηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των κρατικών ε, ενισχύσεων, τι συμβαίνει, δεν ακολουθούν τις δεσμεύσεις που έκαναν, που υπήρχαν οι τράπεζες όσον αφορά το recapitalization ή σε σχέση με μέτρα νομισματικής πολιτικής δεν υπάρχουν υποστηρικτικά μέτρα. Θα ήθελα μία απάντηση και στο φορολογικό ε, τμήμα από πλευρά των κρατών μελών τι συμβαίνει. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά την ποιότητα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την κρατική ε, οικονομία σε σχέση με θέματα δικής σας αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να ε, και για τους λόγους της ε, παρέμβασης είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς αν δεν έχει τις λεπτομέρειες του, τι, το, για το τι γίνεται. Φυσικά δεν μπορούν να ρυθμιστούν τα θέματα της πολιτικής ή να αποκλειστούν ή τουλάχιστον θα πρέπει να μην αναμειγνύονται όσον αφορά την ε, ε, ενίσχυση και την υποστήριξη. Το υπερβάλλον δυναμικό λοιπόν είναι ευλαπτικό. Ποια είναι η αξιολόγησή σας ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δυναμικό της οικονομικής αυτής δράσης, ιδιαίτερα την μέτρηση και αξιολόγηση των κρατικών επιδοτής ενισχύσεων, αν είναι θετικές ή αρνητικές. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια αυτά οι καταναλωτές και ε, μικρή, μικρής κλίμακας εμπλεκόμενοι μπόρεσαν να επωφεληθούν. Τουλάχιστον για την κινητή τηλεφωνία κάνω λόγο για τη χώρα μου και είμαστε γνώμονες για αυτό το αποτέλεσμα. Πολλά όμω σε σχέση με την πολιτική για τον ανταγωνισμό και οι ρυθμίσει που έχουν επιπτώσεις ε, για τους καταναλωτές προέρχονται από του εθνικού ρυθμιστέ. Και εδώ είναι απογοητευτικά τα πράγματα. Είχαμε δύο περιπτώσεις όπου για τον ενεργειακό ρυθμιστή απλά και μόνο υπήρξε τυπική έγκριση για κάποια πράγματα. Και στη συνέχεια όσον αφορά για τον ρυθμιστή των θεμάτων μεταφορών, ρυθμιστική αρχή που βλέπουμε ότι είναι εχθρική για τον ανταγωνισμό η ρύθμιση αυτή και έχουμε και καταδίκη δικαστική που καταδικάζει τον ρυθμιστική αρχή για τις μεταφορές ως ε, ιδιοτελή και ως ε, μεροληπτούντα. Και θα θέλαμε εδώ να το δούμε. Μας ρωτάνε οι καταναλωτές τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Το ερώτημά μου αφορά τις κρατικές ενισχύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία ανήχεται κάνει άνοιγμα στον ανταγωνισμό το α και ω της βιομηχανικής πολιτικής. Πριν από λίγο μιλήσαμε για οικονομική θεωρία. Η οικονομική θεωρία και οι οικονομολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν δραστηριότητες όπου η αγορά υστερεί και που έχει μείνει πίσω και ο ανταγωνισμός είναι αδύνατος, όπως είναι τα φυσικά μονοπόλια, όπως είναι οι δραστηριότητες των δικτύων, μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίε όπου το, το σταθερό κόστος είναι σημαντικό και μια ε, φορολόγηση των περιθωρίων κέρδων ε, ίσως ε, δεν επιτρέψει επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν το κέρδος τους. Οπότε ιδιωτικές επιχειρήσεις εν τη αυτή περιπτώσει μπορεί να μειώνουν την ποιότητα των δικτύων ή όπως διαπιστώνουμε καθημερινά μπορούν να επιβάλλουν πάρα πολύ ψηλά τιμολόγια. Και υπάρχει και κάποια συνεννόηση ολιγοπόλια, φυσικά μονοπόλια που δημιουργούνται στο ιδιωτικό τομέα. Απλούστατο το ερώτημά μου, κυρία Επίτροπε. Θα διευρύνετε το πεδίο των κρατικών ενισχύσεων για να επιτρέψετε κυρίως τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ε, των κοινοφιλών οικονομικών υπηρεσιών. Ή όπως έχουμε και την οικολογική πρόκληση, θα διευρύνετε αυτό το πεδίο ούτως ώστε να μπορούν να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διότι δεν θα εμφανιστούν αυθόρμητα τέτοιου είδους επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Επίτροπε. Η Σωστά έλεγε ότι έχουμε μεγάλη πρόκληση και ότι έχει αναμειχθεί όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτού του είδους την προσέγγιση και ότι συνεργαζόμαστε με την ΕΚΦΙΝ και την, ΕΚΦΙΝ και την Γενική Διεύθυνση την υπεύθυνη για τις αγορές και να δούμε ποια θα είναι η πλήρης πολιτική που θα εφαρμοστεί. Είναι μεγάλη πρόκληση. Και υπάρχουν ειδικέ ομάδες που ασχολούνται. Και είμαι ευγνώμων διότι πριν από λίγο στην αρχή της κρίσης είχαμε επαφές με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με άλλες κεντρικές τράπεζες κρατών μελών για να ζητήσουμε υποστήριξη και να βοηθήσουν με προσωπικό τις ομάδες μας. Χρειαζόμαστε ειδικού αναλυτές, οικονομικούς αναλυτές. Όχι μόνο για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Ακούστηκε κάποιο σχόλιο. Υπόθηκε ότι καμιά φορά υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, αποτυγχάνει η αγορά και πρέπει να το αναλύσουμε το θέμα. Διότι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν έκανε σωστά τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούν, γι' αυτό απέτυχε η αγορά. αλλά με τις συζητήσεις που έγιναν όσον αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες η πρόεδρος υποσχέθηκε ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι στην επόμενη θητεία θα προταθεί πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν. Και αρκετά πράγματα μπορούν να γίνουν. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ποιος κάνει τη δουλειά και ποιος θεσπίζει τα κριτήρια και ποιος διεξάγει τον έλεγχο. Και μιλάμε για τις κοινοφελείς υπηρεσίες που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αναφερθήκαμε στις μεταφορές, στην ενέργεια και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τι λάθη μπορεί να κάνουν αυτές. Θα πρέπει να υπάρχει αναθεώρηση και βαθμολόγηση από ομοτήμους φορείς. Μπορούμε σε διάφορα βήματα να το συζητήσουμε αυτό. Να δούμε τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τι έχουν κάνει σωστά μέχρι τώρα, τι μπορεί να βελτιωθεί. Uh, thank you. Um... Λοιπόν, έχουμε προβλήματα εδώ. Έχω έξι αγόριτες και προτείνω να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις τώρα. Και δεν ξέρω αν η Επίτροπος μπορεί να απαντήσει σε όλες. Ίσως μπορεί να απαντήσει γραπτός, αν δεν έχει χρόνο η Επίτροπος. Τουλάχιστον να ακουστούν όλα τα μέλη. Το Κέπιν, Κάφιν Στήλερ. Είναι τα ονόματα που έχω στον κατάλογο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ερώτηση. Όσον αφορά τα πρόστιμα, είπατε ότι το 2008 επιβάλλατε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ στη Microsoft, αρχές του 2008. Και υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ προστίμου και καταστροφής. Μεταξύ αποτροπής και καταστροφής. Έχει μεγάλη σημασία το ύψος του πρόστιμου. Πώς καθορίζεται το ύψος του προστίμου. Είπατε ότι το όριο είναι 10% του κύκλου εργασιών και καμιά φορά 5% του κύκλου εργασιών. Αλλά τώρα σε αυτή την οικονομική ύφεση 10% του κύκλου εργασιών είναι τεράστιο ποσό που θα πρέπει να καταβάλει σε πρόστιμο μια επιχείρηση. Επίσης, με την καινοτομία. τα πρόστιμα επιβάλλονται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά ή λαμβάνετε υπόψη την καινοτομία της ε, επιχείρησης. Χρειαζόμαστε καινοτομία και θέσει απασχόληση. Όσον αφορά την καινοτομία, η λαμβανεται υποψη την καινοτομια της υστερεί. θεση απασχοληση οσον αφορα ότι πρέπει τα πρόστιμα να λειτουργούν αποτρεπτικά. Δεν θα πρέπει όμω να καταστρέφουν την καινοτομία στην Ευρώπη. Διότι αν τα πρόστιμα έχουν αυτό σαν αποτέλεσμα, τότε αυτοπυροβολούμεθα. Η Κάθριν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Καλές οι κατευθύνες γραμμές για τις ευρωζωνικές υπηρεσίες και η κατάρτιση για τους μειονεκτούντες εργαζόμενους και τους εργαζόμενους με αναπηρία. Πριν από μερικούς μήνες είπατε ότι δεν είναι σύμπτωση ότι τέσσερις από οκτώ τράπεζες με διπλό ε, α σε βαθμολόγηση είναι Αυστραλιανές και εμείς έχουμε μείνει πίσω γιατί ε, ε, μάλλον πάνε καλύτερα ήταν πιο προσεκτικοί. Το αυστραλιανό μοντέλο θα έπρεπε να το στερνιστούμε, πιστεύετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση για αναδιάθρωση του τραπεζικού τομέα. Εκεί, τι απόψεις έχετε για τα προβλήματα του τομέα και ποιοι θεσμοί σας προβληματίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό και στον αμνικό φόρο ε, για τις ε, οικονομικές συναλλαγές. Τι έχετε να πείτε. Σέγε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποια βήματα κατά εκείνων που δημιουργούν καρτέλ. Και 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ έχουν επιβληθεί σαν πρόστιμο. Το υψηλότερο πρόστιμο επευλήθη στην Οβάκη στη Σλοβακία, σε μια χημική βιομηχανία. 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το ποσό είναι πιο ψηλό από αυτό που μπορεί να πληρώσει η επιχείρηση. Και θα μπορούσε να είναι καταστροφικό το πρόστιμο για την επιχείρηση. Μη λησμονείτε παρακαλώ ότι διερχόμαστε κρίση. Στρέφομαι προς εσάς με ένα αίτημα. Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει χρονοδιάγραμμα καταβολής του προστίμου με δόσεις. Η επιχείρηση αυτή είναι σε μια περιοχή όπου υπάρχει ε, μείωση των εργασιών των ορυχείων. Οπότε αυτή η εταιρεία είναι μεγάλος εργοδότης. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν οικονομική καταστροφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Μια παρατήρηση. Μια τάση επικρατεί στην Επιτροπή. Περισσότεροι από εμά, εκτό από εμά που πιστεύουμε στα φυσικά μονοπόλια, θέλουμε να δούμε μια λειτουργούσα αγορά αλλά και εξαιρέσει όταν κινδυνεύουν οι επιχειρήσει. Και τώρα μέσα στην κρίση οι τράπεζε θεωρούνται πολύ μεγάλε για να χρεοκοπήσουν. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον σαν προσέγγιση. Ένα θέμα βρετανικό να θέσω. Η Lloyds TSB και η έρευνα για αυτή την επιχείρηση. Υπάρχουν κάποια πράγματα βέβαια που δεν μπορείτε να πείτε. Τι ερευνάτε όμως μπορείτε να μας πείτε έτσι γενικά. Και ένα από τα θέματα που ερευνώνται είναι το ότι κατά πόσο υπερίσχυσε η Βρετανική κυβέρνηση της αρχής που είναι υπεύθυνη για τα μονοπόλια. Και μήπως μπορείτε να μας πείτε υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήψη απόφασης ε, εκ μέρου σας όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω υποστήριξη προς την ε, Επίτροπο διότι πιστεύω ότι ένας αγώνας κρατικών ενισχύσεων στην Ευρώπη θα ήταν καταστροφικός Είμαι από μικρή χώρα. Και ο κύριος Μπούλμαν προβλέπει κάτι που θα έβλαπτε τη βιομηχανία της χώρας μου. Έχω Saab, Βόλβο στην περιοχή μου, φορτηγά κατασκευάζονται από τη Σκάνια και τη Βόλβο. Και θα μας έβλαπτε αν η Γερμανία μπορούσε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Είμαστε σε ένωση κύριε Μπούλμαν και θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Απευθύνω έκκληση σε εσά, κύριε Επίτροπε να εμείνετε στη θέση σας, να είστε σκληροί. Μόνο έτσι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να επιβιώσει. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιώργη, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εκφράζω την εκτίμησή μου για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε την κρίση και την επενώ για την ευέλικτη προσέγγιση που ήταν χρησιμότατη. Μιλάμε για στατικές εξόδου. Υπάρχει ανάκαμψη σε πολλές χώρες. Θα είναι ασύμετρη η ανάκαμψη. Άλλες χώρες θα ανακάμψουν ταχύτερα και άλλες πιο αργά. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση όταν θα θελήσετε τελικά να καταργήσετε την ευέλικτη προσέγγιση. Απάντηση. Μάλλον η πρόεδρος. Έχουμε ένα πεντάλεπτο, αν κλέψουμε λίγο χρόνο από το επόμενο κομμάτι της συνεδρίασης. Απάντηση. Στα πεταχτά να απαντήσω. Και ζητώ συγγνώμη που δεν θα σας δώσω μια πλήρη εικόνα όσον αφορά κάποια θέματα. Τα υψηλά πρόστιμα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αλλά μόνο έτσι αυτοί που δεν συμπεριφέρονται και δυσκολεύουν τη ζωή των άλλων, τη ζωή των επιχειρήσεων και των καταναλωτών μαθαίνουν το μάθημά τους. Ποια είναι η μέθοδος. Κοιτάμε το, ποιος είναι ο τομέας. Ποια είναι η ζημιά. Ποια είναι η περίοδος κατά την οποία έγινε η ζημιά. Και βέβαια επαναλαμβάνεται αυτή η συμπεριφορά. Τούτων λεχθέντων. Θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχουν πολλές, πολύ περισσότερες επιχειρήσεις που συμπεριφέρονται και συμμορφώνονται από τις άλλες. Καινοτομία, ναι. Αλλά υπάρχουν ένα-δύο παραδείγματα και θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να μπω σε λεπτομέρειε. Αν κάποιο χρησιμοποιεί τη δεσπόρουσα θέση, τότε ο άλλο δεν μπορεί να είναι καινοτόμο. Βλέπετε, μην μιλάτε, μην τονίζετε μόνο την καινοτομία. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμποδίζονται από κακή συμπεριφορά με εταιρείε ή άλλε εταιρείε να είναι καινοτόμε. Θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσει και να αποτρέψουμε τη συμπεριφορά μέσω των προστήμων. Μη δυνατότητα καταβολή του προστήμου, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα συμβαίνουν στην οικονομία εξετάζουμε προσεκτικότατα τις διάφορες επιχειρήσεις και ποια είναι η οικονομική κατάσταση κάθε επιχειρήσης. Τούτου λεχθέντος υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσει κανείς αργότερα και όχι μια δεδομένη στιγμή. Δόσεις από τη στιγμή που θετείται η απόφαση για το πρόστιμο μπορεί να συζητηθεί. Αλλά ξανά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσταλεί το μήνυμα ότι δεν είναι διαφορετική αντιμετώπιση κατά διάρκεια κρίσης από ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Τώρα για τις Αυστραλιανές τράπεζες. Ξέρουμε ότι στο σύστημά τους υπάρχει εποπτεία. και με την προσέγγιση τους ήταν και είναι σε καλύτερη θέση. Και ο κ. Μακρύβη το πρότεινε αυτό στο Κοινοβούλιο. Υπέβαλε κάνα δύο προτάσεις. Δηλαδή να βασιστούμε στα μαθήματα αυτά από την Αυστραλία για το μέλλον. Σλοβακία. Το καρτέλ του... για τουλάχιστον δύο δις ευρώ ζημιά είναι υπεύθυνα τα καρτέλ. Το είπα αυτό. Και όταν δεν μπορούν να πληρώσουν, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πριν επιβληθεί το πρόστιμο, στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλυσε πολύ προσεκτικά την οικονομική θέση της εταιρεία και τη δυνατότητα να πληρώσει. Και συμπέρανε ότι ο αντίκτυπος του προστίμου δεν επηρέαζε μόνιμα τη βιωσιμότητα τη επιχείρηση. Ήξερε η εταιρεία ότι πιθανότατα θα επιβληθεί πρόστιμο και θα μπορούσε να προβλέψει οικονομικά πώ θα το πληρώσει. Το... Όμιλος όμιλο Lloyds Banken. Συμφωνώ ότι μια εύρυθμη αγορά είναι ευλογία για όλους. Για εκείνους που θέλουν δουλειά, για εκείνους που θέλουν βεβαιότητα και ασφάλεια για την οικονομία ο όμιλος Lloyds Banking πράγματι διαμορφώθηκε μέχρι, μέσω εξαγοράς της Halifax, της Bank of Scotland, από την Bank of Scotland μάλλον, και χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από κρατική ενίσχυση που δόθηκε για να σωθεί η Halifax Bank of Scotland. Χρειάστηκαν πολλά χρήματα για την εξαγορά. και αυξήθηκε η παρουσία της τράπεζας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει κρατική ενίσχυση να βοηθάει την τράπεζα να ενισχύσει τη θέση στην αγορά. Γιατί μιλάμε για συγκεντρώσεις εδώ. Δεν πρέπει να είναι εις βάρος των καταναλωτών και των ανταγωνιστών που δεν πήραν ενίσχυση και να χρησιμοποιεί τα χρήματα με τράπεζα για να ισχυροποιήσει τη θέση της. Εξετάζουμε λοιπόν την αναδιάθρωση της Lloyds Bank, το ομίλου Lloyds Bank και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέτρα που έχουν τρεις βασικούς στόχους. Βιωσιμότητα της τράπεζας. Δύο. Επαρκή συνεισφορά της ιδίας της τράπεζας. Και τρίτον, θα πρέπει να είναι ελάχιστο το επίπεδο στρέβλωσης της αγοράς. η σταδιακή κατάργηση της στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Κατά περίπτωση θα εξετάσουμε τη στρατηγική εξόδου και την εκπνοή των μέτρων, τη λήξη των μέτρων. Το είπα και στην αρχή. Δεν θα πρέπει να πειράξουμε τις αρχές μας. Αλλά ο τρόπος εφαρμογής τους θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτος. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό θα κάνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Α, συγγνώμη, ξέχασα μια σημαντική ερώτηση λέει η κυρία Επίτροπος. Όταν μιλάμε για την Όπελ, μόνο εμπορικές πτυχές ελήφθησαν υπόψη, αλλά όπως και με τις τράπεζες. Αν δεν ασχολούμαστε με συγκεκριμένο τμήμα αυτό της αυτοκινητοβιομηχανίας, αν ασχολούμαστε μόνο αυτό, επιβαρύνουμε τους ανταγωνιστές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι λογικό. Όταν πιστεύουμε ότι στο μέλλον χρειαζόμαστε μια πολύ ζωντανή αυτοκινητοβιομηχανία και θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία να ενισχυρεί η αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και είναι ίσως και το σωστό μήνυμα αυτό για, να, για την τελευταία παρέμβασή σε αυτή την Επιτροπή. Σε ευχαριστώ που ήρθατε και σε ευχαριστώ και τις άλλες φορές που ήρθατε για να μας μιλήσετε και να μας ενημερώσετε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τώρα. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Στέρξ όσον αφορά τις αιτήσιους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εταιριών όσον αφορά τις μικρομονάδες. Όσοι ε, κινείστε παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία και όσοι θέλουν να συζητήσουν να σπάνε έξω από την αίθουσα γιατί γίνεται θόρυβος και δύσκολο να μιλήσει ο κύριος Στέρξ. Σας ευχαριστώ. Ντέρκ, λυπάμαι που σε πίεσα χρονικά, αλλά έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Έχουμε μία πρόταση τη ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μην ε, ε, ε, εγκαταλείψουν την ε, ε, την ιδέα των ετησίων λογαριασμών για τις μικρές μονάδες. Δεν πιστεύω όμως ότι η πρόταση που αποβλέπει σε μία εξαίρεση για τις μικρές αυτές ε, επιθέσεις επιχειρήσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κανείς τη γραφειοκρατία και πιστεύω ότι έχει πολλά μειονεκτήματα διότι πρέπει να θυμηθείτε ότι όταν μιλάμε για χρηματοδότηση για μικρές μονάδες αν δεν υπάρχει διαφάνεια πώς θα προχωρήσετε εάν ε, θέλετε να υπάρξει χρηματοδότηση εφόσον θα χρειαστεί να παρουσιάσετε ε, ορισμένους λογαριασμούς δηλαδή ε, θα, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα. Επίσης θα πρέπει να έχετε ένα, μια ισότιμη ε, αντιμετώπιση ε, διότι ε, διαφορετικά Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα ε, στο οποίο ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία. Υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες ε, στον τομέα αυτό σε διάφορες χώρες όπως η δικιά μου και τότε θα ήταν πολύ καλύτερα να υπάρξει μια χωριστή κατηγορία επ' αυτού διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε και ε, θα ε, δούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσουμε ε, τις επιχειρήσεις και να δούμε εάν μπορούν να να παρουσιάσουν ε, καλύτερα τα αποτελέσματά τους. Θα πέριπτα λοιπόν την πρόταση αυτή και θα ζητούσα από την Επιτροπή του χρόνου να εξετάσει χωριστά το θέμα των μικρών επιχειρήσεων, να μειώσει το διοικητικό βάρος με μια αναδιάρθρωση της τετάρτης οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Φιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. οι υποχρεώσεις ετησίων λογαριασμών για τις μικρομονάδες οδηγούν σε μία σύγκρουση συμφερόντων διότι ε, καταρχήν ε, υπάρχει μία μία ανισορροπία μεταξύ των βαρών και ε, των υποχρεώσεων. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να έχετε μία σαφή εικόνα της επιχειρήσεως, να μπορέσετε να εντοπίσετε ποιες είναι οι φορολογικές της ανάγκες ε, ε, φορολογικές υποχρεώσεις και όλα αυτά να γίνονται με τρόπο διαφανή. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις ε, εθνικές ε, συνθήκες σε μία περίοδο κρίσεως και να μπορέσουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να εξασκήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες με έναν τρόπο εναρμονισμένο και συνεκτικό. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του διασυνοριακού εμπορίου και οι κανόνες που διατυπώνουμε να είναι συγκρίσιμοι. Ένα απλοποιημένο σύστημα ετησίων λογαριασμών για τις μικροεπιχειρήσεις είναι μεν αναγκαίο και επιθυμητό διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφανθεί στο θέμα αυτό το 2008 και πρέπει να λάβουμε υπόψη της μικροεπιχειρήσεις οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται μόνο σε μία χώρα ή μόνο σε μία περιφέρεια ή επαρχία και να δούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν ε, επηρεάζουν ε, γενικώ την οικονομία της χώρας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι τις Ιουνίου ήμουν επικεφαλής ε, μιας επιχειρήσεως σε μια ισχυρή οικονομική περιφέρεια της Γερμανίας και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη μειώσεως ε, γραφειοκρατίας και το ότι όλοι λέγουν ε, ότι χρειάζεται μικρότερη, λιγότερη γραφειοκρατία αλλά επειδή ήμουν επικεφαλής μιας επιχειρήσεως μεγάλης αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται να υποβάλλονται ορισμένα στοιχεία. Όταν λοιπόν βλέπω τι έχει υποβάλει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η η πρόταση αυτή ε, μειώνει και τις πληροφορίες που δίνονται και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε ε, πώς τα κράτη-μέλη ε, διαφοροποιήσουν ε, τις ε, υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων από τις μικρές τους επιχειρήσεις ε, για να έχουν και στατιστικά στοιχεία και ε, μία φορολογική εικόνα. Οπότε εάν δεν έχει επαρκέσει η έρευνα που έγινε, αν δεν ξέρει κανείς πώς θα επηρεάσει η νομοθεσία αυτή τις μικρές επιχειρήσεις και αν θα υπάρξει όντως μία μείωση της επιβαρύνσεως ε, για τις μικρές επιχειρήσεις ή ε, αν τελικά σε εθνικό επίπεδο η γραφειοκρατία αυτή οδηγήσει σε ίσως και μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Ε, γι' αυτό θέλω να παρακολουθήσω και να συμφωνήσω με αυτά τα οποία ζητά ο κύριος Στέρξ και ιδίως ότι πρέπει να γίνει μία εκτενής έρευνα κατά τρόπον ώστε ε, το 2010 όταν θα υπάρξει μία ε, αναδιαπραγμάτευση της 4 και της 7 οδηγίας τα στοιχεία αυτά να ληφθούν υπόψη. Έχω ακόμη πέντε θα παρακαλούσα λοιπόν να είστε σύντομος. Ο πρώτος είναι ο Ζων Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τις αναλύσεις που έγιναν και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο θέμα αυτό υπήρξε μία συζήτηση σύμφωνα με αυτά που είπε ε, που είπε ο εισηγητής μας για το ότι έγινε πέρυσι. Ενδέχεται λοιπόν η αναδιάρθρωση αυτή τελικά να είναι αρνητική αλλά πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο είχε ε, δράσει πολύ σοφά. Είχαμε πει ότι άμεσα καταρχήν πρέπει να υπάρχουν απαλλαγές και ε, διευκολύνσεις για τις εταιρείες που δεν έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες και η Ευρώπη θα πρέπει να προτείνει με ένα πιο απλοποιημένο σύστημα ε, λογιστικής παρουσιάσεως των ε, στοιχείων για τις μικροεπιχειρήσεις. Ε, βέβαια το να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ αυτής της αλλαγής με την αναδιάρθρωση της, ε, των σχετικών οδηγιών θα ήταν προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων και όχι εις βάρος τους. Η κυρία Κιούρη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. αν, αν υιοθετηθεί αυτή η οδηγία ως έχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία θα σημαίνει 95% από αυτές δεν θα έπρεπε, δεν θα χρειάζεται να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς και διατάξεις όσον αφορά του αιτήσιους απολογισμού, λογιστικούς απολογισμού, πράγμα το οποίο θα είχε αρνητική επίπτωση. Γιατί θα έπρεπε ειδικέ εκθέσεις να συνταθούν για να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει ε, των ουγγρικών διατάξεων. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Θα πρότεινα να μην υιοθετήσουμε ως έχει αυτό το κείμενο. Τώρα, αν επιχειρήσεις ε, υπό την οροφή και υπό τις διατάξεις που προβλέπονται από το σχέδιο οδηγίας θα έπρεπε να μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες οι εταιρείες τι θα κάνουν αν θα εφαρμόζουν την απλουστε, τους απλουστευμένους κανονισμούς ή όχι. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να ξαναδούμε και να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό των οροφών και αυτών των πλαισίων, γιατί θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό σε κάποιες χώρες. Ο κύριος Λάγκεν παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να ξανααναφερθώ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Όμως τον Δεκέμβριο 2008, όχι τόσο παλιά, δηλαδή στο παρελθόν, στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίσαμε οι μικρές επιχειρήσεις να ανακουφίζονται, να απαλλάσσονται από τα στατιστικά αυτά στοιχεία. Τώρα εξελέγει νέο Κοινοβούλιο, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Τα επιχειρήματα όμως που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν εξακολουθούν να ισχύουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν διατάξεις για τις μικρές, μικρότατες αυτές επιχειρήσεις, αλλά να δούμε αν θα εντάσσονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν αφορούν την μια εσωτερική αγορά. Δεν δραστηριοποιούνται διασυνοριακά αλλά μόνο τοπικά. Και γι' αυτό δεν χρειάζονται ευρωπαϊκοί κανονισμοί και διατάξει για αυτέ τι μικρότατε, μικρών διαστάσεων επιχειρήσει. Εμεί γνωμοδότηση πρέπει να δώσουμε σε Ευρωκοινοβούλιο. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ουσία. Είναι απόλυτα λάθο, απόλυτα λανθασμένο μια και μια μεγάλη υψηλών. Ε, αξιωματούχων ομάδα ασχολήθηκε με τη μείωση της γραφειοκρατίας και του γραφειοκρατικού βάρους, εδώ να επιβαρύνουμε τις μικρότατες επιχειρήσεις με ε, γραφειοκρατικό άχθος. Όπως τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστά τα πράγματα. Μπορεί να συζητήσει κανείς για προθεσμίες, διορίες και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά τώρα όπως το συνιστά ο κύριος Τάξ να απορριφθεί είναι βελγική πολιτική και όχι ευρωπαϊκή. Γι' αυτό απορρίπτω αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Um, Οι δύο τελευταίοι αγορητές, Πιτ Κάνιν και μετά Βόρτμαν Κόλ, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Επειδή αναφέρθηκαν πολλά και υποστηρίζω απόλυτα την προσέγγιση του κυρίου Στέξ στην πρότασή του ουσιαστικά θα έλεγα μεγάλη βλάβη θα γινόταν για τις επιχειρήσεις και για τις ίδιες τις μικρές επιχειρήσεις, για την κοινωνία, τους καταναλωτές και τους ευρωπαίους καταναλωτές αν δεν είχαμε συμφωνήσει κανονισμούς και διατάξεις που θα εφαρμόζονται για αυτούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ, σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την Επιτροπή Μεταφορών, ο κύριος, κύριε συμφωνώ μαζί σας με την πρόταση σας. Όμως αυτήν εδώ την πρόταση που έχουμε μπροστά μας δεν μπορώ να συμφωνήσω πάντα επανειλημμένα επαναλαμβάναμε ότι μικρέ και μικρότερε επιχειρήσει πρέπει να ανακουφιστούν από το γραφειοκρατικό βάρο. Τώρα υποβάλλει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ούτε καν την εξετάζεται με σοβαρό τρόπο. Την απορρίπτεται συλλήβδην και λέτε ε, του χρόνου, ίσω την επόμενη χρονιά μπορεί κάτι να γίνει. Όχι λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή σήμερα πρέπει να υποστηριχθούν οι μικρέ και μικρότερε επιχειρήσει. Φυσικά μπορεί η πρόταση αυτή ίσω να προσαρμοστεί. Όμω στη δική σα έκθεση πάτε πολύ βιαστικά για την απόρριψη. Κύριε Στέρξ, θέλετε να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προσέξτε, κύριε Λάγκεν. Δεν γνωρίζω αν γνωρίζετε καλά Ολλανδικά για να με καταλαβαίνετε όταν ομιλώ Ολλανδικά. Φαίνεται ότι δεν με προσέχετε, αλλά τέλο πάντων αν θεωρείτε ότι ακολουθώ βελγική πολιτική εδώ, τότε πρέπει να σα απαντήσω εσεί ακολουθείτε γερμανική πολιτική και όχι ευρωπαϊκή πολιτική. Α μην χρησιμοποιούμε λοιπόν τέτοια επιχειρήματα. Οι αμφιβολίε μου λοιπόν δεν αναφέρονται στο ότι αν τώρα είναι αναγκαία η γραφειοκρατική ανακούφιση και ελάφρυνση ή όχι. Το ερώτημα είναι, αυτή η πρόταση είναι η σωστή οδός ώστε για τις μικρότερες, επιχειρήσει επιχειρήσεις να υπάρξει απλούστευση και ανακούφιση. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Φαίνεται ότι ίσως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Φαινομενικά. Τα φαινόμενα πατούν όμως. Κάποιοι συνάδελφοι το είπαν. Κάποιες απαιτήσει ε, δεν εξαλείφονται τελείως στη, λέτε ότι δεν υπάρχουν ε, μικρότατε επιχειρήσεις που να ασχολούνται διασυνοριακά όμω στη χώρα μου συμβαίνει αυτό και ο Πορτογάλος συνάδελφος το ανέφερε για αυτού του είδους επιχειρήσεις λοιπόν διοικητικά θα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα επειδή πολύ λιγότερο θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα άλλων επιχειρήσεων. Και τότε είναι δύσκολο λοιπόν, πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει χρηματοδότηση για αυτές τις επιχειρήσεις, διότι εξακολουθούν οι, τράπεζες να απαιτούν θέματα διαφάνειας, διαφάνεια. Εδώ έχουμε απαιτήσει στατιστικές, ε, απαιτήσει σε σχέση με, τη, με δεδομένα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι στις περισσότερες χώρες στατιστικά δεδομένα διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο θα συλλέγονται αυτό τι είναι, απλούστευση, είναι ανακούφιση γραφειοκρατική. Δεν είναι σαφέ αυτό, διότι θα πρέπει πάλι να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία και πληροφορίε. Πάλι θα πρέπει να συμπληρώνουν έντυπα και τέτοιου είδου ε, αιτήσει ε, ή ε, να συναλλάσσονται με αυτόν τον τρόπο επιχειρήσει. Εδώ θα πρέπει να δοθεί μια κατεύθυνση ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθηθεί για την ανακούφιση και απλούστευση στην αναθεώρηση της οδηγίας και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει γοργά. Δεν πρόκειται λοιπόν για την επιβάρυνση που θέλουμε να διατηρηθεί, γραφειοκρατική επιβάρυνση ή να αυξηθεί, αλλά δεν είναι το, ο σωστός τρόπος αυτός να το πετύχουμε εδώ. Είμαι πρόθυμος να συζητήσουμε για τροπολογίες με συναδέφους, ώστε στο τέλος τέλος να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να ε, παρέμβουν και πάλι. όμω ο συντάκτη γνωμοδότησης θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσω θα μπορούσε κανεί να εξετάσει αυτή την πρότασή του, όπω την ανέφερε, για να υπάρξουν κάποιε τροπολογίε που θα ικανοποιήσουν και θα λύσουν το πρόβλημα. Η προθεσμία διορία για τι τροπολογίε θα είναι η 2η Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι οι κοινοβουλευτικέ ομάδε έχουν ήδη ειδοποιηθεί ότι μόνο αγγλικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα τροπολογιών, γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβουμε τι ψηφοφορίε στην Επιτροπή Αρμόδια τη Ουσία. Τροπολογίε μέχρι τι 2 Οκτωβρίου, το 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στι 6 Οκτωβρίου αυτές τις τροπολογίες. Σας είδα κύριε Λάγκεν, ζητείτε τον λόγο. Σας λέω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό βρισκόμαστε υπό αυτή την χρονική πίεση. 6 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εμείς στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην Επιτροπή Αρμόδια Επιτροπή 10 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί. Θα καταλήξουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και μπορούμε ίσως ε, να προλάβουμε και να προσαρμόσουμε και εμείς τις εργασίες μας. Το θέμα θα ήταν αν χάσουμε αυτές τις ημερομηνίες θα ε, έχει νόημα να συντάξουμε γνωμοδότηση. Λάγεν, διαδικαστικό πρόεδρε. Αν και αγγλικά είναι η μητρική σα γλώσσα, δεν θέλουμε εδώ να εισαγάγουμε νέου κανόνε, έτσι δεν είναι. Μέχρι σήμερα μόνο στα αγγλικά μιλούσαμε και συντάσαμε τροπολογίε όταν πρόκειται για την ένταξη νέων μελών στην Ευρωζώνη. Και παρακαλώ αυτό ο κανόνα ε, για, για έναν Ευρωβουλευτή που θα έχει δικαίωμα να έχει όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να ψηφίσει στη μητρική του γλώσσα να είναι σεβαστό και στο μέλλον όταν έχουμε Βρετανό στην Προεδρία ή Αγγλόφωνο. Παρακαλώ και να ζητήσετε να παρατηρήσετε παραταθούν οι προθεσμίες για την ψήφιση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αν είναι αναγκαίο. Το θεωρώ απαραίτητο να μπορέσουμε να σεβαστούμε αυτού τους κανόνες στην αρχή τη κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ. Κύριε Λάγκεν, Έχω μεγάλη κατανόηση και συμπάθεια για αυτά που λέτε. Όμω, ωστόσο, δεν πιστεύω ότι συσχετίζεται η απέτηση για τα αγγλικά με μένα ω Προεδρεύουσα. Είναι κάτι που το κάναμε και στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία για να επιταχύνουμε τα πράγματα. Μια κοινή γλώσσα που κατανοούν οι περισσότεροι. Σημείωσα αυτό που είπατε. Να ζητήσουμε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη ουσία να παρατείνει τι διορίε. Το θέμα είναι <clears throat> αν δεν γίνεται, οι τροπολογίε δεν γίνονται δεκτέ στα αγγλικά και οι συντονιστέ ε, είχαν ειδοποιηθεί ικανοποιηθεί, κανένας δεν είχε διατυπώσει κάποια ένσταση. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την απέτηση, έχουμε την εναλλακτική λύση ε, για τη γνωμοδότηση που πώς θα πετύχει. Δεν έχουν ζητήσει, δεν έχει αναφερθεί τίποτα από τους συντονιστές ω παλαιά συντονίστρια θα ήθελα να υποστηρίξω το αίτημα του κ. Λάγκεν και να ζητήσω και οι άλλε γλώσσε να χρησιμοποιηθούν. Παρακαλώ τα γερμανικά, σίγουρα τα γαλλικά, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω έχθρα κατά των Αγγλικών, αλλά μετά από πέντε χρόνια εμπειρία τι διαπιστώνω ότι πάντα πιεζόμαστε από τι προθεσμίε και στην πραγματικότητα μετά περνάει πολλή χρόνο μέχρι να περάσει το κείμενο. Ήμουν εισηγητή για δύο μεγάλα χαρτοφυλάκια, με πίεσαν, το έκανα και μετά πέρασαν 6-7 μήνε πριν οι, γλω... νομικοί να κάνουν τη δουλειά του. Εγώ έκανα στο νοσοκομείο στα δυτική θητεία μου, είμαι δικηγόρο. Και με έμαθαν ότι δεν υπάρχουν κατεπήγοντα στα νοσοκομεία παρά μόνο διαστικοί άνθρωποι. Αν δεν υπάρχουν κατεπήγοντα στα νοσοκομεία και εδώ το κατεπήγον του πράγματο πρέπει να είναι σχετικό. Κοιτάξτε, αν τα μέλη θέλουν να υποβάλουν σε άλλε γλώσσε πέρα των Αγγλικών, και αν οι μεταφράσεις δεν είναι στη διάθεσή μας μπορούμε να αναβάλουμε τη συζήτηση και ψηφοφορία και αν δεν το κάνει η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή δεν θα υπάρξει γνωμοδότηση και εκεί τελειώνουμε. Μπορώ να κάνω τα δέοντα διαβήματα. Κύριε Στέρξ, θέλετε το λόγο. Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να εργαστώ στα αγγλικά κυρία Πρόεδρε. Εάν όμως επιτρέψετε γαλλικά και γερμανικά υπάρχουν και μερικές άλλες εγώ δεν έχω πρόβλημα να εργαστώ στα αγγλικά. Αλλά βέβαια τίθεται και θέμα αρχή. Αν οι συντονιστέ πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν γνωμοδότηση. Αν δεν υπάρξει γνωμοδότηση, τελικά ίσως να είναι κρίμα. Πρόεδρος, ο... εάν δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα να τηρήσουμε προθεσμία, θα πρέπει να δεχθούμε ό,τι υποβάλλουν τα μέλη. Άρα τα αφήνω στη διακριτική ευχέρεια των μελών. Μπορούν να υποβάλουν στην γλώσσα τους άλλες γλώσσες. Δεν βλέπω άλλη λύση. Πήρα απόφαση. Η απόφαση είναι ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι το μεσημέρι στις 2 Οκτωβρίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σας ή τη γλώσσα κάποιου άλλου και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εάν δεν καταφέρουμε να επιβραδύνουμε την καθήλια αρμόδια επιτροπή και αν δεν έχουμε έτοιμες μεταφράσεις, αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Τα μέλη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σύμφωνα με αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα Νόμιζα ότι πέρασε η στιγμή του ενθουσιασμού. Όμως μας περιμένουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ζων Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρο της Ευρωομάδας. Παρακαλώ, αν θέλετε να συζητήσετε καθηδίαν, βγείτε έξω. Οι συζητήσεις να γίνουν εκτός εθούσης της Επιτροπής. Η τελευταία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιούνκερ έγινε στις 31 Μαρτίου 2009. Βεβαίω θα έχουμε τη δυνατότητα και για άλλη ανταλλαγή απόψεων. Το 2010 δεν συμφωνήσαμε συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά γίνονται τακτικέ συναντήσει. Θα ακολουθήσουμε παρόμοια μορφή που συνηθίζουμε. Θα γίνει μια παρουσίαση στον κύριο Γιούνκερ, που μετά θα ακούσει τι ερωτήσει σα. Έχετε το λόγο, λοιπόν, κύριε Γιούνκερ. Κυρία Πρόεδρε, πραγματική χαρά για μένα να αντιπροσωπεύσω στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή σας, να εκπροσωπήσω την ομάδα μου και διπλή χαρά μου διότι βλέπω και την κυρία που προεδρεύει τη Επιτροπής που είναι πολύ σημαντική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σας. Την τελευταία φορά που παρουσιάστηκα μπροστά σας ήταν τέλος Μαρτίου ενεστώτος έτους και σε εκείνο το ραντεβού η οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης όπως την περιέγραψα ήταν κακή. Διαπιστώνω ότι η οικονομική κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κατά πολύ και στην κοινή γνώμη επικρατεί μια μέτρια αισιοδοξία όσον αφορά το δεύτερο εξάμεινο ενεστώτος έτους και για όλο το έτος 2010. Όμως θα ήθελα και εγώ να εκφραστώ με μεγάλη, με, συνε, με συνετή προσέγγιση. Η κυρία Λούλινγκ Κυρία Λούλινγκ, καθίστε παρακαλώ. Γιατί αυτή η συνετή προσέγγιση και η μετριοπάθεια. Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά το μέγεθος ανάκαμψης και το ρυθμό της ανάκαμψης. Είναι έφραστη οικονομική κατάσταση. Και δεν έχουμε δικαίωμα από την άλλη να δημιουργήσουμε ψευδείς προσδοκίες διότι η κρίση από την οποία βγαίνουμε σταδιακά ήταν βαθιά κρίση και οι συνέπειες των βαθέων κρίσεων γίνονται αισθητές επί μακρά περίοδο. Και όσον αφορά τα δημοσιονομικά, τις χρηματοστρικές αγορές και την απασχόληση του των λεχθέντων. Θεωρώ όμως ότι βγήκαμε από την ελεύθερη πτώση της οικονομίας της Ευρωζώνης και το καταφέραμε το πρώτο εξάμεινο ενεστώτος έτους. Έχουμε μια πραγματική σταθεροποίηση. Από το φθινόπωρο του 2008 η πολιτική δράση περιορίστηκε ουσιαστικά στη διαχείριση της κρίσης. Απρόβλεπτα γεγονότα μας υποχρέωσαν στη θέσπιση εκτάκτων μέτρων εκτός του πλαισίου αναφοράς του θεωρητικού. Καταπολεμήσαμε τη φωτιά με φωτιά και συμφωνήσαμε ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή. Όμως, συμφωνούμε λέγοντας ότι αυτά τα μέτρα δεν ήταν μόνο έκτακτα, αλλά έπρεπε να έχουν και προσωρινό χαρακτήρα και θα έπρεπε να εφαρμοστούν στατηγικές διεξόδου από τη στιγμή που θα επέτρεπε κάτι η κατάσταση, ώστε να αποφύγουμε το να γίνουν τα δημοσιονομικά πολύ έθραυστα και να αυξηθούν οι στρεβλώσεις που θα, θα προκαλούνται από τα έκτακτα μέτρα. Υπήρξε συμφωνία σχεδόν γενική Μάλιστα αυτό παγιώθηκε και από τους G20 στο Pittsburgh. Πρέπει να επικαιροποιηθούν αυτές οι στρατηγικές εξόδου ούτως ώστε να είναι λειτουργικές και να εφαρμοστούν τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι έχουμε μια γερή ανάκαμψη. Όμως υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρονική στιγμή που θα είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες εξόδου από την κρίση η οικονομική και χρηματοδοτιστική κατάσταση και οι βραχυπρόθεσμες μεσοπρόθεσμες προπτικές συζητούνται στις συνεδριάσεις του Eurogroup και τους ECOFIN, ECOFIN αυτής της Πέμπτης και Παρασκευής και σε τι συνεδρίσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου εναστότος έτους, 2009, το 2009 θα χαρακτηριστεί από μεγάλη μείωση του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάπτυξη ήταν πολύ αρνητική το 2009, 4%. Πρέπει να επενθυμίσω ότι αυτή η σταθεροποίηση της καταστάσεως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εθελοντικές δράσεις των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων. Όσον αφορά το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα βασιστούν σε μια μέτρη ανάκαμψη της δραστηριότητας της τάξης 0,3%-0,5%. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω κάτι που τίνουμε να λησμονούμε στις ανοιχτές συζητήσεις και στη δική μας συζήτηση και επελήφθη του θέματος η Ευρωμάδα, το Eurogroup, τις προπτικές ανάκαμψης. Ποια ανάκαμψη μπορεί, θα μπορούσε να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας πλήρως παραγωγικές δυνατότητες χωρίς να δημιουργήσουμε πληθωρισμό μεγάλο. Αποδεικνύεται ότι ότι η δυνατότητα ανάπτυξης στην Ευρωζώνη λόγω της κρίσης ε, θα μειωθεί αρκετά. Έχουμε δυνατότητα, είχαμε μικρή δυνατότητα ανάπτυξης, 2,5% και φαίνεται τώρα δεδομένο μετά την κρίση ότι θα στρέφεται η ανάπτυξη κοντά στο 1,5% για την περίοδο 2010-2020, δυνατότητα ανάπτυξης η συζήτηση όσον αφορά τη θεωρητική ανάπτυξη έχει σημασία διότι αυτή η θεωρητική ανάπτυξη, μέτρια θεωρητική ανάπτυξη συνάδει με μέτρια οικονομική δραστηριότητα και περιορίζεται το δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών για τους πολιτικούς ε, φορείς. Εντός της Eurogroup προσπαθούμε να ε, αναζωογονήσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική συλλογική και να φροντίσουμε ο καθένας να κάνει το καθήκον του στο σπίτι του. Έχοντας υπόψη μας ότι τα διαθροτικά ταμεία με συγκεκριμένους στόχους θα οδηγήσουν σε καλύτερη ανάπτυξη και σε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση. Αυτή η συζήτηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης, για τις προπτικές ανάπτυξης είναι σημαντική όχι μόνο λόγω των διασυνδέσεων με τη συζήτηση για τη στρατηγική εξόδου από την κρίση, αλλά επειδή δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να δώσουμε νέα όθηση σε, διαθωτικές, σε σχήματα για να αναζωογονήσουμε την ανάκαμψη. Η κατάσταση λοιπόν σταθεροποιήθηκε και μπορούμε να δούμε έναν ε, σχετικά ρόδινο ορίζοντα. Λοιπόν, η κρίση πώς επηρεάζει την ανάπτυξη των χωρών μας, το είπαμε αυτό. Έχουμε άλλα δύο θέματα που να εξετάσουμε και εξετάζουμε στην Eurogroup η ανάπτυξη και τι γίνεται με τα δημοσιονομικά, ποια είναι η κατάσταση των δημοσιονομικών. Εγώ εξετάζω, έχω πάντα υπόψη μου την κοινωνική διάσταση Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θέλω να είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα. Πάντα έχω στην καρδιά μου αυτό το θέμα και η ανάπτυξη που θα γνωρίσουμε τους επόμενους μήνες στην αγορά εργασίας θλίβει και ανησυχεί. Βλέπουμε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, είδαμε στους πρώτους τρεις μήνες, ότι λόγω μείωση οικονομικής δραστηριότητας θα αυξηθούν οι απώλειες θέσεων εργασίας και αρκετοί πολίτες μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται πιέσεις για να βρουν ε, λύσεις. Εξού και η σημασία του θέματος της θεωρητικής δυνατότητας ανάπτυξης που προανέφερα, το δυναμικού ανάπτυξης. Η αύξηση ανεργίας θα έχει κακές κοινωνικές συνέπειες για αυτούς που πλήττονται και τι τις οικογένειές τους, πέρα από τα προσωπικά δράματα θα υπάρξει και αύξηση φόρτου των δημοσιονομικών που θα πρέπει να πούμε ότι ήδη αντιμετωπίζουν ακραίες πιέσεις. Θα υπάρξει διαθροτική ανεργία που είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Το βλέπουμε ήδη. Αυτό έχει συνέπειες στην εμπιστοσύνη και τη συμπεριφορά των οικοκυριών και των καταναλωτών. Την εμπιστοσύνη όμως τη χρειαζόμαστε, ούτω ώστε η κατανάλωση να συνεχίζει να τροφοδοτεί την οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε διτό στόχο. Να αποφύγουμε τις απολύσεις στο μέγιστο δυνατό και μεσοπρόθεσμα να γίνει πιο ισχυρή δομή των οικονομιών μας, ούτω ώστε να αντισταθούν καλύτερα στους κλονισμούς. Τρίτη, μέρημνα η κατάσταση των δημοσιονομικών. τελευταίους 12 μήνες μελετήσαμε το θέμα. Έγιναν προσπάθειες, σταθεροποιήθηκαν οι οικονομίες μας. Και τα έκτακτα μέτρα όμως που μας βοήθησαν δεν μπορούν μέσω μακροπρόθεσμα να παραμείνουν. Πρέπει ήδη να σκεφτούμε ποια θα είναι η στατηγική εξόδου από την κρίση και κυρίως για την Ευρωζώνη διότι έχουμε κοινό νόμισμα. Ξεκινήσαμε στη Eurogroup όπως και στο ΕΚΟΦΗΝ, να εξετάζουμε από κοινού ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η στρατηγική εξόδου. Πρέπει να συντονίσουμε τα βιολιά μας, αν θέλετε, τις προσπάθειές μας και να δούμε τι αλληλεπίδραση έχουν τα διάφορα μέτρα υποστήριξης και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την κατάργηση των μέτρων, των εκτάκτων. Και αυτά στο πλαίσιο Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όταν εφαρμόστηκε αυτό το σύμφωνο, δεν προβλέψαμε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση που γνωρίζουμε σήμερα. Ευτυχώς η μεταρρύθμιση που κάναμε τον Μάρτιο του 2005 μας έδωσε περισσότερα περιθώρια να κινηθούμε. Μπορέσαμε να εφαρμόσουμε ευέλικτα τα μέτρα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτή η ευελιξία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευελιξία που δεν είναι αμφίδρομη. Χρειάζεται να καθεριωθούν διαδρομές εγγύσεις σταθεροποίησης και στόχοι φιλόδοξοι. Η εφαρμογή με εξόδου δεν μπορεί να εφαρμοστεί τώρα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα. Δεν ήρθε η ώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα design, ένα σχεδιασμό στρατηγικών εξόδου αλλά δεν φτάσαμε σε τέτοια ορίμανση της σταθεροποίηση για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Το 2010 δεν θα είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής στρατηγικής διεξόδου, αλλά από το 2011 και μετά σταδιακά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή για την έξοδο γνωρίζοντας βέβαια ότι προφανώς δεν μπορούμε να αρκεστούμε όσον αφορά τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών σε μικρά βήματα. Η σταθεροποίηση και η μείωση των ιδιωτικών ελλημάτων θα, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι έχουμε τέτοια ελλείμματα πάνω από το 0,5% ε, το χρόνο που είχαμε προβλέψει δεν μπορούμε να εξετάζουμε μεμονωμένα τη στατηγική εξόδου, τη δημοσιονομική. Η Ευρωμάδα, το Eurogroup, θέλει να, να έχει γενική στρατηγική εξόδου, συντονισμένη στρατηγική εξόδου. Αυτή η στατηγική θα συμπεριλαμβάνει τα κάτωθη στοιχεία. Επιστροφή των δημοσιονομικών σε μια πορεία βιωσιμότητας υποστήριξη, μεταρρύθμιση διαθροτική χρειάζεται για να βελτιωθεί η ανάπτυξη και θα πρέπει οι χρηματοδοτικέ αγορές να επιστρέψουν μια χρηματοδότηση άνευ υποστήριξη. Ο καλός συντονισμό του στρατηγικών εξόδου είναι πάρα πολύ σημαντικός και σε διεθνέ επίπεδο και εντό της Ευρωζώνης και είναι προφανέ ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδράσεις μεταξύ των διαφόρων μέτρων που ελήφθησαν για να εξασφαλίζεται η οικονομική και η χρηματοστική σταθερότητα. Εξίσου φανερό είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαδράσεις όταν θα συζητήσουμε την λήξη εφαρμογής αυτών των μέτρων. Και το χρονοδιάγραμμα πάυσεως αυτών των μέτρων θα εξαρτάται κατά χώρα, από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να δούμε όλα τα προβλήματα που τίθεται χωρίς να έχουμε ταμπού και να γίνει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων. Κάτι που προέβλεψαν οι συνθήκες. Το Eurogroup όπως και το ECOFIN θα πρέπει να σεβαστούν την κατανομή των αρμοδιοτήτων και το καθεστώς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε στο σύνολο τους τα προβλήματα. Χρειάζεται ευρεία θεώρηση των προβλημάτων παρά μια στενή θεώρηση στρατηγικών εξόδου στο δημοσιονομικό τομέα. Να πω και κάτι κυρία Πρόεδρε όσον αφορά τους G20. Η Eurogroup υποστηρίζει τη θέση υποστήριξε η Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου και η ομάδα G20 όσον αφορά τις στρατηγικές εξόδου που απαριθμούνται στην τελική ανακοίνωση και όπως η αρχιτεκτονική προτείνεται για το χρηματοδοτικό τομέα στο διεθνές επίπεδο και υποστήριξη επίσης των φτωχών χωρών που πλήττονται πιο σκληρά από την κρίση από ότι οι ευρωπαϊκές χώρες. Οι G20 καθόρισαν το πλαίσιο για τις συζητήσεις που αφορούν την μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της δίκης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ξεκίνησε συζήτηση όσον αφορά τις διάφορες ομάδες G, που έχουν δημιουργηθεί, G7, G8, G14, G20, G20 που έχει περισσότερα μέλη από το 20 που αναφέρει ο τίτλος G20. Το κοινοβούλιο σας πάντα υποστήριζε την Ευρωμάδα και πάντα ζητούσε εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης που θα είναι ισχυρή, συμπαγής, συνεκτική έχοντας υπόψη την οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Ούτω ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε αποτελεσματικά με τους ομολόγους μας τους διεθνείς, τα οικονομικά θέματα πώς. Οι ανισορροπίες που υπάρχουν, ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών και τις ισοτιμίες του ευρώ. Θα πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία που μας δίνει η συζήτηση για την διακυβέρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να έχουμε μία εκπροσώπηση στο εξωτερικό της Ευρωζώνης που να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, στις διεθνείς φιλοδοξίες και να συνάδει με το καθεστώς του ενίου νομίσματος που είναι το δεύτερο ε, διεθνές ε, νόμισμα και περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις που θα έχετε την καλοσύνη να μου υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Έχουμε ως πάντα εντυπωσιακό αριθμό μελών που θέλουν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αν θέλετε με τον Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω πολύ σύντομες ερωτήσεις. Στο νέο κόσμο, μετά την στρατηγική διεξόδου 2011, αν άκουσα καλά όπως αναφέρατε, θα βρεθούμε σε ένα κόσμο μη συγχρονισμένο θα υπάρχουν χώρες που θα μπορούν να βρουν διέξοδο από την κρίση νωρίτερα, κάποιες άλλες που πολύ αργότερα θα εξέλθουν από την κρίση. λαμβάνοντα υπόψη εκείνες που θα φύγουν πιο νωρίς από την ε, κρίση, είναι οι κυριότερε χώρες υπό οικονομικού όρου Και μετά από την παρέμβαση του κυρίου Τρισέ εχθέ μπορεί να δημιουργηθεί μια νομισματική στρατηγική διεξόδου με την αύξηση των ε, επιτοκίων όταν θα έχει παγιωθεί η ανάκαμψη. Και εδώ πάλι θα έχουμε, ας το πω έτσι, για τις πιο καθυστερημένες χώρες ε, ε, την τη μάστιγα. Δεν θα είναι λοιπόν ενιαία αυτή η στρατηγική. Θα είναι μεταβλητής γεωμετρία στρατηγική ανάλογα με τι διάφορε χώρε. Επίση, κατανόησα ότι πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών. Αλλά για τι πιο καθυστερημένε χώρε ε, αυτό θα είναι δυνατόν όταν θα υπάρξει ενδυνάμωση τη ε, ανάπτυξη. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Ερώτησή μου για μετά την Λισαβόνα εποχή. Θεωρείτε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη περίοδο πέρα από τα 10 χρόνια λαμβάνοντα υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μεγαλύτερη εμβέλεια. Το πρόβλημα του ανταγωνισμού ήταν ένα πρόβλημα για την Ευρώπη πριν και μετά από την κρίση. Η υπεργύρανση δημογραφική και κυρίω η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού θεωρείται ότι επαρκούσε, ήταν επαρκή. Ή μήπω αυτή η έλλειψη δυνατοτήτων να υπάρξουν επιλύσει στο πρόβλημα εξηγεί εν μέρη την αποτυχία τη στρατηγική ε, τη προσέγγιση Λισαβόνα. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να ενισχυθεί η ελλειψη δυνατοτητων να υπαρξουν λυσει στο προβλημα εξηγει εν μερη την αποτυχια τη στρατηγικη τη προσεγγιση λισαβονα γι αυτο θα ηταν σκοπιμο λοιπον να ενισχυθει η κυβέρνηση, αν γίνεται. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε να υπάρξει μια πραγματική διπλωματία του ευρώ με μια φωνή και ενία πολιτική. Όμω το στοιχείο κλειδί είναι η μεταρρύθμιση και κυρίω η μέθοδο, ώστε οι συστάσει τη Ευρωομάδα ουσιαστικά να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη και να συμμορφωθούν. Ευχαριστώ. We'll try θα προσπαθήσουμε ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση, αν συμφωνείτε. Αν όμως καθυστερήσουμε θα παίρνουμε ομάδες ερωτώντων. Νομίζω ότι η στρατηγική για να βγούμε από την κρίση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί αναλόγως της χώρας. Δηλαδή τα κράτη της Ευρωζώνης δεν βρίσκονται όλα στην ίδια κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι η ίδια από τη μια χώρα στην άλλη και ε, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ο οποίος θα είναι συντονισμένος για να δούμε ποιος θα είναι ο ρυθμός που θα υιοθετηθεί από κάθε χώρα για να υπάρξει μία διέξοδος ε, από την ε, κρίση όσον αφορά το πρόγραμμα της Λισαβόνας που δεν αναφέρεται μόνο στην ε, Ευρωζώνη αλλά σε 27 κράτη-μέλη εγώ παρόλο που δεν είμαι εξιοδοτημένος ε, μπορώ να σας πω ότι θα ήθελα προσωπικά να παρατείνουμε την περίοδο αναφοράς θεωρούμε ότι η αρχική περίοδος αναφοράς ε, μέχρι το 2010 δεν μπορεί πλέον να ισχύσει και θα έπρεπε να ε, να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε μέχρι το 2020 χωρίς όμως κατά αυτόν τον τρόπο να ε, επιβραδύνουμε τις τις μεταρρυθμίσεις αλλά πιστεύω ότι αυτό το πλαίσιο αναφοράς το ισχύον δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί. Τι χρειάζεται ε, για να εφαρμόσουμε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, χρειάζεται η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού δεν λέω όχι δεν θεωρώ ότι η μέθοδος αυτή καλύπτει όλα τα στοιχεία μιας ενδιαφέρουσας προσέγγισης αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες κατά τρόπον ώστε ορισμένες κυβερνήσεις να δώσουν μια ενισχυμένη ε, δυνατότητα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε, στην Ευρώπη και ε, καλύτερα θα ήταν ε, να, αντί να δίνουμε προθεσμία στις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις ε, να ε, αντιδράσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουν υπερβολική Ευρώπη. Για μένα πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι αυτή που χρειαζόμαστε αλλά χρειάζεται ακόμη ένα βήμα το οποίο εγώ μένει με έτοιμος να κάνω όχι όμως οι υπόλοιποι όλοι. Ο κύριος Μπόμαν. Κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, εν ονόματι των Σοσιαλιστών και Δημοκράτων σας καλωσορίζω στο νέο Κοινοβούλιο. Έχει κάπως αλλάξει οι ονομασίες πολιτικής μας ομάδας γιατί στην Ιταλία δεν έχουμε ε, μόνο σοσιαλιστές αλλά σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες και φιλελεύθεροι οι οποίοι έχουν ε, διαφορετική προσέγγιση προς την Ευρώπη. Απλώς διευκρινίζω δηλαδή και έχω δύο ερωτήσεις οι οποίες έχουν ε, στενή σχέση με τις προηγούμενες. Δηλαδή, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωομάδα ε, ε, είναι ε, όταν θα υπάρξει η δεύτερη συνθήκη της Λισαβόνας θυμάστε τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια αλλά θα πρέπει στην Ευρωομάδα να γίνει μία συζήτηση για να δούμε τις διάφορες διαστάσεις της στρατηγικής πολιτικής και να να εξετάσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι κατεπήγον. Δεν θέλουμε να είμαστε μονοχρωματικοί. Δεν θέλουμε δηλαδή να βρεθούμε ε, αποκλειστικά σε μια στρατηγική, η οποία θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και η οποία θα αμφισβητεί τις άλλες πολιτικές μας. Επίσης ε, στη συζήτηση του Πίτσμπαρκ πριν και μετά ζητήσαμε για μια συνολική οικονομική διακυβέρνηση ε, και είπαμε ότι καλό είναι να υπάρχει λογική διακυβέρνηση διεθνώς αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην Ευρωζώνη δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα ή στην Ευρώπη δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα και αυτή είναι η διαφοροποίησή μου στη συζήτηση ρωτώ λοιπόν εσείς πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο των Ευρωπαίων σε μια τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να τεθούμε στο περιθώριο και θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή μας πολιτική, να μπορέσουμε να εκφραζόμαστε με μία φωνή, διότι θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με ε, την φορολογία των ε, οικονομικών ε, συναλλαγών καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα. Ξέρετε ότι είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά με τους σοσιαλιστές εγώ αισθάνομαι πάντοτε καλά, ατυχώς μειώνεται συνέχεια έχει ο ρυθμός των σοσιαλιστών. Οπότε θα ήθελα να, να αυξηθούν για να αισθάνομαι ακόμη καλύτερα όσον αφορά τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρες και εγώ είμαι της γνώμης ότι όπως κάναμε και στο Λουξεμβούργο το 2005 ε, ολοκληρώσαμε την ατζέντα της Λισαβόνας με τις πολιτικές διαρθρωτικές αλλαγές και με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κατά τρόπον ώστε ε, να υπάρχει καλύτερη κοινωνική συνοχή διότι θεωρώ ότι ε, είναι μία σωστή ανησυχία και ε, έχει σημασία για την ατζέντα της Λισαβόνας. Ένα θέμα μας λείπει ακόμη. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας υπερτιμήθηκε και η κοινή δράση για περιβαλλοντολογία λογική, πολιτική έχει υποτιμηθεί ενώ πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να συζητούνται στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Έχει σημασία όλα αυτά να μπορέσουν να έχουν καλή έκβαση και θα πρέπει να, να ασχοληθούμε με, τα, όλα τα βασικά μας συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η επίπτωση της οικονομικής κρίσης, γενικότερης κρίσεως, ε, θα πρέπει να μην ε, ε, οδηγήσει σε ε, μία αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας ή στην παραμέληση ορισμένων διαστάσεών της. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ΕΚΟΦΗΝ, Ευρωπαϊκού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ούτω καθεξής, πιστεύω ότι η στους G20 υπάρχει η επιθυμία η ομάδα G20 να αποτελέσει μία παγκόσμια κυβέρνηση σε οικονομικά θέματα και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός των οικονομικών μέτρων αλλά θα πρέπει θα πρέπει στην ομάδα αυτή να καλύπτεται το 90% του ΑΕΠ θα πρέπει οι ευρωπαϊκές θέσεις να καταρτίζονται σωστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο ΕΚΟΦΗΝ κατά τρόπον ώστε οι Ευρωπαίοι οι οποίοι συμμετέχουν στο G20 να αισθάνονται ότι είναι δεσμευμένοι από την εντολή που έχουν λάβει από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους πράγμα το, από το οποίο αποκλίνουν στις συνεδριάσεις τώρα και γι' αυτό αποδυναμώνουν τη θέση τους. Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, δεν πρέπει να γίνει μια γενική γραμματεία του G20. Υπάρχουν 192 ε, ε, μέλη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οπότε δεν μπορεί ε, οι 20 του G20 απλώς να κατανείμουν τις αρμοδιότητες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος που ζητά το λόγο είναι η Σιλβί Γκουλότ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω σχετικά με την εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ. Δηλαδή να εκφράσουμε την ε, ίδια ανησυχία ότι ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα υπόκειται στους G20. Σε αυτό μου απαντήσατε. Αλλά τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα μετά την ε, ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είπατε δεν προηγουμένως ότι θέλετε να ξεπεράσουμε, ε, να υπερβούμε την ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Ε, αντιλαμβάνομαι την κόπωσή σας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε στους ψηφοφόρους και να τους πούμε το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί διότι καταρτήθηκε το 2000 όπου υπήρχαν 15 εκατομμύρια άνεργοι. Άρα τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να μας βοηθήσει στον τομέα αυτό. Για να ξεκινήσω την απάντησή μου θα βασιστώ στο δεύτερο στοιχείο της ερώτησής σας σχετικά με την ατζέντα της Λισαβόνας. Ήθελα να σας πω ότι ίσως δεν με καταλάβατε σωστά. Η ιδέα μου δεν είναι να ε, πετάξω στα σκουπίδια την ατζέντα της Λισαβόνας, απλούστατα, να υπάρξει ένα ε, πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Δηλαδή το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να περιέχει ημερομηνίες οι οποίες θα μπορούν να υπερβαίνουν το 2010 που ήταν η αρχική ημερομηνία που είχαμε προβλέψει σαν τελική προθεσμία όταν υιοθετήσαμε την συνθήκη της Λισαβόνας υπό την, την ατζέντα της Λισαβόνας υπό την προεδρία του κυρίου Γκουτιέρης αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να είμαστε όμως πιο ρεαλιστικοί γιατί είπαμε ότι μέχρι το 2010 θα πρέπει θα πρέπει να ε, μην σταματήσουμε άρα ρεαλιστικά θα πρέπει ε, να ε, παρατείνουμε τις προθεσμίες χωρίς να επιβραδύνουμε τις ημερομηνίες εφαρμογής των διαφόρων στοιχείων της Λισαβόνας. Επίσης όσον αναφορά τις υπόλοιπες διεθνείς οργανώσεις σαν G20 και άλλοι η Ευρώπη θα πρέπει ε, να ε, παρουσιάζεται με τη τάλα τη στοιχεία ε, Ευρωζώνη και τα λοιπά. Ξέρετε ότι υπάρχει μία συζήτηση σχετικά με τις δικαιοδοσίες που δεν συζητείται τώρα τόσο ισχυρά διότι ορισμένοι είχαν πιέσει την Ευρώπη και η μόνη οποίοι θέλουν να μειώσουν τα μέλη από 24 σε 20 ε, ε, ε, πετώντας έξω ορισμένους Ευρωπαίους είναι οι Αμερικανοί και θέλουν επίσης να αποκλείσουν ορισμένες αναδιόμενες χώρες οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της παγκοσμίου οικονομίας. Δεν νομίζω θα το πετύχουν διότι η μείωση των ε, συστατικών μελών ε, δεν ε, είναι μία συζήτηση η οποία έχει λήξει. Είμαι όμως ο ίσως ο τελευταίος των Μοϊκανών που ζητά να υπάρχει μία θέση για την Ευρωζώνη, μάλλον είμαστε δύο και ζητούμε ε, το ίδιο να υπάρχει και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο, παρόλο που δεν ενθουσιάστηκαν ε, στην Ευρω... Ε, στο Ευρωγκρουπ όταν προτόλμησα να προτείνω μία τέτοια λύση η οποία βέβαια δεν έτυχε χειροκροτήματος διότι ακόμη και στην Ευρωζώνη ε, η κάθε, κάθε χώρα ε, έχει μία ισότεμη θέση ε, ενώ πιστεύω ότι αν συγκεντρώναμε όλες τις προσπάθειές μας σε μία έδρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ήμασταν πιο αποτελεσματικό αλλά αυτό θα γίνει ίσως σε κάποιον άλλο αιώνα. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούνκερ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε εδώ μετά από το κομματικό συνέδριό μας όπου <clears throat> υπήρξε αυτή η επίσκεψη και κυρίως θα είχα μία ερώτηση προς εμάς. Αναφέρεται στην ερώτηση των απολογισμών και των μη ισορροπιών στην Ευρωζώνη. Δεδομένης της διαφοράς των μισθών παρέκκλησης μισθών και μισθολογικών δαπανών και των πλεονασμάτων πριν από την κρίση της Γερμανίας μέσα στην Ευρωζώνη απολογισμού σχετικός. Σας ερωτώ, ποια είναι τα μέτρα ουσιαστικά, ποια είναι, ποιες είναι οι συγκεκριμένες επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης για την ε, σταθερότητα του ευρώ που μεσοπρόθεσμα μπορεί να διακυβευτεί, θεωρώ. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι απλά οι χώρες εκείνες που έχουν ε, ελλείμματα πρέπει να μειώσουν προς τα κάτω, λέει, του να προσαρμόσουν προς τα κάτω τους μισθούς τους. Ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά είναι εφικτό αυτό. Το να καταλήξουμε σε μια κατάσταση αποπληθωρισμού είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Ερώτηση, ποια μέτρα λοιπόν μέσα στην ευρωομάδα εξετάζονται συγκεκριμένα για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ποιε επιπτώσει πρέπει να συνεπάγεται αυτό για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Δεν πρέπει να συμπληρωθεί με μια εξωτερική διάσταση αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Διότι αυτή η παρέκκληση που σημειώνεται όσον αφορά τους απολογισμούς θα πρέπει να αποφευθεί. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την προσωπική σας τοποθέτηση επ' αυτού, αλλά και τι τοποθετήσει μέσα στην Ευρωζώνη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η ερώτησή σα: Τουλάχιστον 17 απαντήσεις μπορεί να δοθούν σε αυτήν την ερώτηση. Για κάθε χώρα εσωτερικά και ξεχωριστά θα πρέπει κανεί να αναφέρει τι κάνει η κάθε κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και πώς τα εκτιμά. Τώρα, όσον αφορά τις εσωτερικές μη ισόρροπες σχέσεις, αυτό το θεωρώ σαν κάτι που δεν ε, διακυβεύει, δεν, δεν δημιουργεί κίνδυνο υπαρξιακό για το ευρώ. Όμως είναι κάτι που συνολικά έτυχε ε, ελλειπούς προσοχής μέχρι τώρα. Και μέσα στον κύκλο των Υπουργών της Ευρωζώνης συμφωνούμε όλοι ότι συστημικά, συστηματικότερα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με πιο στοχοθετημένη αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου των παρεκκλήσεων και διαφορών και της ε, αποκατάστασης των ισορροπιών σε περίπτωση μετάθεσης ή αποσταθεροποίησης. Πρέπει να απασχοληθούμε περισσότερο σε βάθος με αυτό. Αυτές οι μη ισόρροπες σχέσεις ε, που υφίστανται αλλά που δεν δημιουργούν κίνδυνο αποσύνθεσης ή ε, κίνδυνο διακύβευσης του ευρώ διότι υπάρχουν και αλλού τέτοιου είδους παρεκκλήσεις δεν υπάρχει κάποιος τύφλος ούρτης ή κάποια οδηγία από πλευρά της Ευρωομάδας για τη μείωση αυτών των μη ισόρροπων αναλογιών. Παρότι σταθερά με αργό ρυθμό κινούμαστε προς, ε, κάποιο τέτοιο στόχο, προς ένα τέτοιο στόχο. Δεν υπάρχει όμως ακόμα κάποια οδηγία όμως εξετάζεται σε τακτά διαστήματα και υπάρχει η έμονη, η ιδέα και η έντονη ιδέα από πλευράς ε, χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ότι όταν υπάρχουν παρεκκλήσεις ε, από τη γενική γραμμή κάποιων χωρών θα πρέπει εκείνοι που παρεκκλίνουν να θέσουν εντάξει τα του οίκου τους. Εδώ είναι θέμα, ας το πω έτσι, της ε, διευθέτησης από πλευράς της Ευρωζώνης των παρεκκλήσεων και έχουμε και τα αιτήματα αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και να επανορθωθεί. Και αυτό κάνουμε, αυτό βρισκόμαστε καθοδόν να κάνουμε, ώστε τέτοιου είδους μη σώροπες σχέσεις και δυσαναλογίες να μην επεκταθούν και δημιουργούν κίνδυνο. Κατά τα άλλα, υπάρχει και κάποια, ας το πω έτσι, ε, αντίσταση, ε, δημιουργεί ένα είδος ε, αλλεργίας να υπάρξει τέτοιου είδους υποβάθμιση ή επικριτική αντιμετώπιση της ζώνης ευρώ υπάρχει έντονη ε, έκκληση από πλευράς των ΗΠΑ προς την Γερμανία ώστε να, υπάρξει συνεισφορά από πλευράς της ε, Γερμανίας ώστε να επανορθωθούν οι ε, μη ισόρροπες σχέσεις και δυσαναλογίες. Η Ευρωζώνη όμως διεθνώς δεν μπορεί να το δεχθεί να κατακαιρματίζεται. Οι άλλοι παρακαλώ, οι εκτός Ευρωζώνης πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη Ευρωζώνη και πρέπει ως Ευρωζώνη να αντιμετωπίζεται και όχι με κατακαιρματισμένο τρόπο διαχωριστικά ως Γερμανία ή ε, ξεχωριστές ε, χώρες ε, για την αποκατάσταση ισορροπιών. Κατά τα άλλα για την Ευρωζώνη σε σχέση με ένα ε, σύνολο δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα για την ε, ύπαρξη των μη ισόρροπων σχέσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι σε σχέση με την Ευρωζώνη μια συγκεκριμένη τέτοια τοποθέτηση θα πρέπει πάντα να αποβαίνει προς την αποκατάσταση των μη ισόρροπων σχέσεων. Και κατά τα άλλα ε, θυμάμαι με ευχαρίστηση το συνέδριο σε, σχέση με τον κύριο Μπούλμαν όμως τι ήταν το πρασίνο σε σχέση με την S5 όμως φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει τέτοια πρόσκληση λυπούμε γι' αυτό σας ευχαριστώ κύριος Γκέμπερ Ευχαριστώ πρόεδρε ο πρόεδρος Γιούνκερ μόλις μας είπε ότι θα παραμείνει ασαφές το οικονομικό παγκόσμιο περιβάλλον και χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια διακυβέρνηση οικονομικά. Το G20 κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το μέλημα διότι το G20 είναι μία κατά περίπτωση ε, συγκρότηση χωρίς ε, σαφείς κανονισμούς, χωρίς νομική βάση και δεν εξαρτάται από το σύστημα των ε, Ηνωμένων Εθνών. Όντως το G20 είναι ε, μία επιστροφή στα συνέδρια των ε, μεγάλων δυνάμεων, συνέδριο της ε, Βιέννης ή περιπτώσεις όπου ορισμένες χώρες σαν την Ιταλία ή τη Γαλλία θέλουν να κυβερνήσουν τον υπόλοιπο χρόνο. Υπάρχουν όμως δημοκρατίες σαν την ε, ε, Σαουδική Αραβία στο G20 οπότε δεν θέλω αυτοί να με διευθύνουν. Οπότε κύριε Γιούνκερ εσείς είπατε ότι το G20 ε, δίδει οδηγίες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή άλλους οργανισμούς που έχουν τους ίδιους κανόνες τους. Δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε να αντικατασταθεί το G20 στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών από ένα οικονομικό συμβούλιο ασφαλείας για να παραμείνουν όλα αυτά στα πλαίσια του διεθνούς ε, δικαίου. Συμφωνώ ως προς την ανάλυση. Άλλωστε σας είπα σε μία παρέμβαση ότι ε, δεν θα ήθελα να ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ε, υπόκειται στο G20 διότι πιστεύω ότι η ιδέα ε, της G20 δεν είναι κακή διότι χρειαστήκαμε στην αρχή και κατά τη διάρκεια της κρίσεως περισσότερη και καλύτερη διαβούλευση από ό,τι στο παρελθόν. Το G20 όμως πρέπει να σκεφτεί ε, πώς θα διαμορφώσει την εσωτερική του διάρθρωση. Δεν υπάρχει ούτε γραμματεία ούτε έδρα. Αυτό θα ε, ε, εξαρτηθεί από τους G20 και από τους Ευρωπαίους να αποφασίσουν και να οργανωθούν κατά τρόπον ώστε ε, οι συντεταγμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάζονται σωστά στο G20 και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή, στην διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για ένα νέο θέμα δεν πρόκειται για νέο θέμα, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από καιρού καιρών και θα έπρεπε να τοποθετηθεί σωστά στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όλοι. Εγώ δεν θα ήθελα να με διοικήσει η Γενική Συνέλευση των ε, Ηνωμένων Εθνών διότι εκεί η Σαουδική Αραβία δεν είναι απομονωμένη λόγω της κατακριτέας ε, θέσης της σχετικά με τη δημοκρατία. Στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν πολλές μη δημοκρατίες οπότε ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, θυμάστε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ε, βέτο <laughs> για ορισμένους προνομιούχους. Αντιθέτως ε, συμφωνώ μαζί σας κατά εν μέρη ότι υπάρχει κίνδυνος το G20 να γίνει ε, ένα παιχνίδι μεγάλων δυνάμεων σαν τον 19ο ε, ή τις αρχές του 20ου αιώνα διαγράφεται ένας τέτοιο κίνδυνος χωρίς όμως να έχουμε αυτή τη στιγμή τους ίδιους κανόνες όπως υπήρχαν στο 19ο αιώνα. Ε, το παιχνίδι αυτό ξεκινάει από τον 19ο ε, αιώνα και γι' αυτό δεν μιλώ για τον 20ο ή τον 21ο, όπου είναι πιο πολύμορφο το παιχνίδι. Ε, ε, ε, θα μπορούσα να απαντήσω σε γλώσσα του Λουξεμβούργου στον κύριο Γκέμπελς κατόπιν των σχολείων τα οποία έγιναν προηγουμένως. Νομίζω ότι το γλωσσικό το λύσαμε, θα σας πω μετά. Ο επόμενος που ζητά το λόγο είναι ο κύριος Γιούργεν Κλούτ. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούγκερ, είπατε ήδη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την αγορά εργασίας. Εγώ προέρχομαι από τη Γερμανία όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εκλογές και προεκλογικό αγώνα. Η ανεργία για μας ε, θα αυξηθεί πολύ τους επόμενους μήνες και η κρίση κατά δεν έχει μετριαστεί όπως είπατε στην αρχή. Πρόκειται για κλιμακώσεις και πιστεύω ότι όσον αφορά την αγορά εργασίας τα προβλήματα είναι μπροστά μας και δεν είδα να λεχθούν τόσα πολλά στο Πίτσμπεργκ για το πόσο θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς σαν Ευρωγκρουπ τι, τι συγκεκριμένες προτάσεις έχετε προς τους συμμετέχοντες κατά τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα πληγούν εντός των επομένων μηνών να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν της οικονομικής πολιτικής διότι όπως είπατε πολλοί πολίτες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα άρα δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους τους γιατί είδαμε εις τις ευρωεκλογές ότι η συμμετοχή μειώνεται συνέχεια διότι οι πολίτες ε, αναρωτιόνται τι εποφελούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε πρέπει να τους διευκρινίσουμε ότι και οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες σαν εργαζόμενοι μπορούν κάτι να περιμένουν να έχουν κάτι στο οποίο προσβλέπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εντύπωσή μου είναι ότι σε αυτά τα οποία είπα εισαγωγικά ότι η παγκόσμια οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν βρίσκονται πλέον σε ελεύθερη πτώση το θέμα της ανεργίας και της αγοράς εργασίας και της υποαπασχόλησης όμως θα μας χτυπήσει, θα μας πλήξει με μεγάλη ένταση στο άμεσο μέλλον. Μπορεί κανείς να πει ότι τους επόμενους μήνες σε σχέση και με το έτος 2010 στη συνέχεια και μετά το 2011 θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Το ποσοστό των ανέργων στην Ευρώπη δραματικά θα αυξηθεί και σύμφωνα με τον παλαιό γνωστό εμπειρικό κανόνα ότι μια κρίση στην αγορά εργασίας φτάνει και ολοκληρώνεται και με δραματικές διαστάσεις όταν έχει, όταν έχει σταθεροποιηθεί ε, η, οικονομία και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και θα το δούμε ότι και στην Ευρωζώνη η ανεργία βρίσκεται εντωμεταξύ στο 9,5% ως ποσοστό. Αυξήθηκε, μια και βρισκόταν κάτω από 7% αυτό το ποσοστό στο παρελθόν κατά τα πρώτα έτη της ε, ύπαρξης ε, του κοινού νομίσματος. Τα πρώτα δέκα χρόνια λοιπόν της ύπαρξης του ευρώ η ανεργία μειώθηκε, εντάξει. Και πολύ συχνά έχουμε ουσιαστικά την απόδειξη που προσπαθήσαμε να δώσουμε ότι η ανεργία θα έτεινε προς τα κάτω επειδή υπήρχε το ευρώ και υπήρχε η πειθαρχική, ας το πω έτσι, επιβολή, η τάση επιβολής της πειθαρχίας. Έγινε αυτό. Τώρα πρέπει να μεριμνήσουμε για άλλη πειθαρχία, άλλου είδους πειθαρχία σε σχέση με την Ευρωζώνη να υπάρξει συμμόρφωση ώστε αν όχι αμέσως στο εγγύς μέλλον να υπάρξει σταθεροποίηση πάλι των αγορών εργασίας. Γι' αυτό πιστεύω έντονα ότι δεν ήρθε τώρα, δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή ώστε τα πακέτα οικονομικής ανάπτυξης να τερματιστούν ξαφνικά. Δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ οπωσδήποτε ότι τα δημόσια οικονομικά, τα οικονομικά, ο, οικονομικός ο κόσμος της οικονομίας με μια επεκτατική δημοσιονομική τάση και το 2009 και το 2010 χρειαζόμαστε μια διευρυμένη δημοσιονομική πολιτική. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε στραγγαλιστικά να την τερματίσουμε αυτή την πολιτική και πρέπει συντονισμένα να δράσουμε για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι διατάξεις ε, οι προδιαγραφές ε, μερικής απασχόλησης όπως υφίστανται θα πρέπει να συνεχιστούν. Και αυτό θα έχει ως επίπτωση τα δημόσια οικονομικά να, ε, να να επιβαρυνθούν και τώρα έχουμε, αν όποιος θέλει να οδηγήσει στην άμεση λήξη των διατάξεων προσωρινής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης θα επιβαρύνει κατά πολύ και θα πλήξει την οικονομία σίγουρα. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε το δυναμικό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη να ενδυναμωθεί και σε σχέση με το 5% που βρισκόταν πριν από την κρίση αυτό το δυναμικό για το επόμενο δεκαετές διάστημα θα είναι στο 1,5% πράγμα το οποίο σίγουρα δεν επαρκεί ως ε, ποσοστό ανάπτυξης ώστε οι αγορές εργασίας ε, να ισορροπηθούν. Γι' αυτό πρέπει στις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις δεν μ' αρέσει πάρα πολύ ο όρο προσαρμογέ και μεταρρυθμίσει, διότι κάθε ένα κατανοεί ότι επιθυμεί υπό αυτό. Και η ατζέντα τη Λισαβόνα, αν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα, θα καταρρεύσει. Και γι' αυτό δεν θέλω να εκτεθούμε σε αυτόν τον κίνδυνο. Παρότι υφίσταται αυτό ο κίνδυνο, πάσης φύσεως μέτρα απορρίθμισης ε, ή ε, χαλάρωσης που ε, στην πρακτική πολιτική ε, προτείνονται δεν θεωρώ ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Δεν πιστεύω ότι η λήξη, η εκπνοή των ρυθμίσεων για τις απολύσεις ε, θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Το αντίθετο κιόλας. Υπάρχει ο κίνδυνος χωρίς προστασία έναντι των απολύσεων με την μείωση του επίπεδου προστασίας των εργαζομένων να καταλήξουμε σε κύματα απολύσεων και σε μέγα πρόβλημα ανεργίας. Καταδείχθηκε ότι σε σχέση με είπαν κάποιοι ότι αν υπήρχε λήξη εκπνοή των διατάξεων για την, τις απολύσεις θα οδηγούμαστε σε ανάκαμψη. Τέτοιου είδους αφελείς προβλέψεις και προσδοκίες δεν με βρίσκουν σύμφωνο και γι' αυτό θα πρέπει μέσα στην Ευρωζώνη να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προστατευτούμε. Ευχαριστώ. Κύριο Σκυλακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αναδείξατε την κρισιμότητα των διαθροτικών αλλαγών. Ταυτόχρονα όμως μιλήσατε για μια παράταση ρεαλιστική της ατζέντα της Λισαβόνας κατά μία δεκαετία η πρόθεση των διαθροτικών αλλαγών ασφαλώς δυσχεραίνεται από την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χρηματοδοτήσει κανείς τις μεταβατικές περιόδους και γενικότερα τις διαθροτικές αλλαγές με πολύ κακά δημόσια οικονομικά. Ταυτόχρονα μιλήσατε για έναν χαμηλό μεσοχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης, 1,5% που ασφαλώς δεν είναι αρκετός για να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο πακέτο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Ένωση, ένα συνδυασμό κοινωνικών πολιτικών, κλιματικών αλλαγών και σταδιακής βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την υπόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών νωρίτερα ενδεχομένως, ήδη από το 2010 μαζί με τον σταδιακό σχεδιασμό για τον περιορισμό των ελλημάτων ως πότε θα αναβάλουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρέπει να επιμείνω και να αντιδράσω λέγοντας ότι δεν ζητώ να σταματήσει η εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων της ατζέντα της Λισαβόνας. θα κάνω μία έκκληση για παράταση της προθεσμίας μέσα στην οποία θα μπορέσουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των ε, μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της ατζέντα της Λισαβόνας. Εγώ λοιπόν δεν ξέρω πότε πρέπει να ξεκινήσουν οι, οι διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει να συνεχιστούν. Έχουν γίνει πολλές ε, δομικές ε, μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, άλλες επέτυχαν, άλλες όχι, άρα δεν πρέπει να ξεκινήσουμε αλλά να συνεχίσουμε χωρίς να υπάρχει καμία στάση και οι κυβερνήσεις είναι προσιλωμένες σε αυτή την ατζέντα της Λισαβόνας. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα το οποίο αναφέρεται εις ε, τη στρατηγική δημοσιονομικής ε, διεξόδου την οποία αναφέρατε και όπως σας είπα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ε, αποσύρουμε τα δημοσιονομικά κίνητρα από την οικονομία αγοράς μας δηλαδή δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική πολιτική την οποία έχουμε εφαρμόσει με αρκετή επιτυχία. Το 2010 ε, δεν θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμοστεί μία τέτοια στρατηγική. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε για το πώς θα διαρθρωθεί και θα διαμορφωθεί η στρατηγική διεξόδου. Και γιατί. Διότι πιστεύω ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα έκτακτα προσωρινά μέτρα τα οποία έχουμε περιλάβει στο σύστημα δεν θα, δεν θα ισχύσουν για πάντα ότι έχουμε επιβαρύνει τους προπολογισμούς μας και οι νέοι επομίζονται αυτή τη στιγμή το βάρος των πολιτικών που εφαρμόζουμε τώρα και που πρέπει να εφαρμόσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Αλλά για να έχει εμπιστοσύνη ο καταναλωτής και να μπορέσει να βλέπει την άκρη του τούνελ θα πρέπει ε, να, να διατυπώσουμε μία στρατηγική που θα επιτρέψει να ε, εξέλθουμε από την επιβάρυνση των ελλημάτων και να υπάρχει μία στρατηγική διεξόδου η οποία θα διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί από κοινού. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν ε, μία μέρα να αποφασίσει ο Γάλλος Πρωθυπουργός ότι τέρμα ε, ή η καγκελάριος της Γερμανίας θα αποφασίσει να συνεχίσει ή κάποιος θα αποφασίσει ε, να τελειώσει με την, να αποπληρώσει τα χρέη τον Ιούλιο παραδείγματος χάνει και οι άλλοι θα συνεχίσουν να κομμαχάνε θα πρέπει να υπάρχει μία στρατηγική διεξόδου από τα δημοσιονομικά προβλήματα και τα μη συμβατικά μέσα που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει ε, να ισχύσουν. Σεβόμαστε την ε, ανεξαρτησία της τραπέζης αλλά όλα τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν νομισματικά, δημοσιονομικά, πολιτικά και άλλα είναι συνδεδεμένα ε, Κύριε Γιούγκερ, θα πάτε ε, στο Γκότενμπεργκ όπου ε, θα συναντήσετε τον κύριο Μπορντέλ και τον ε, κύριο Μπόργκ που παρουσίασαν προεβδομάδων εβδομάδων το πρόγραμμα. Ο κύριος Μπόργκ λοιπόν μας είπε ότι δεν είναι βέβαιος ότι ήταν καλό ότι ήταν εκτός της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Εσείς είσαστε πιο βέβαιος για τις επιπτώσεις όσον αφορά τον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Ορντέλ ο οποίος είπε ότι ήταν προσόν για τη Σουηδία ότι ε, δεν ήταν ε, στην Ευρωζώνη διότι είχε πιο αδύναμο νόμισμα και μπόρεσε να αυξήσει τις εξαγωγές της. Τι πιστεύετε λοιπόν κύριε Γιόνκερ και ρωτώ διότι πρέπει να υπάρξουν ε, σοβαρές συζητήσεις με τους ε, δύο Σουηδούς ομολόγους σας για να έχετε καλά επιχειρήματα για την σημασία του ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ιδίω, καθότι θα χρειαστούν επιχειρήματα για να πείσουν τη Σουηδική κοινή γνώμη ότι το ευρώ είναι καλό πράγμα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τη Σουηδία και σας εύχομαι καλό ταξίδι. Ε, εφόσον βέβαια είμαι Πρωθυπουργό στο Λουξεμβούργο. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή την ε, διακυβερνητική διαμάχη μεταξύ ε, Σουηδίας και άλλων δηλαδή συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Μπόργκ διότι πολλές φορές όταν συζητούσαμε αυτό το θέμα ε, ξέφρασα τη γνώμη ότι σύμφωνα με την αντίληψη και την ε, πεποίθησή μου η ε, Ευρώπη της Σουηδίας είναι μέσα στο ευρώ, δεν υπάρχει λόγος να παραμένει έξω και αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Όταν λοιπόν θα πάω να τους επισκεφτώ θα τους πω ότι έχουμε την ίδια γνώμη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα να επανέλθω στο δημόσιο έλλειμμα που αναφέρατε, που είναι αβάσταχτο. Υπάρχουν τρει τρόποι να μειωθούν αυτά τα ελλείμματα. Να μειωθούν οι δαπάνες, να αυξηθούν οι φόροι και να αυξηθεί η ανάπτυξη. Όταν αναφέρατε την ε, διαθετική μεταρρύθμιση θα πρέπει φαντάζομαι να μειωθούν κάποιες δαπάνες. Τι σκέφτεσαι για την αύξηση των φόρων και κυρίως κάποιους φόρους που όλο και λιγότερο βαρύνουν το κεφάλαιο και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ήθελα να ξέρω με αυτή την προοπτική μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων των κρατών τι σκέφτεστε όσον αφορά μια φορολόγηση των οικονομικών χρηματοστικών συναλλαγών, την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, αύξηση των φόρων όσον αφορά τι εταιρείε που μειώθηκε κατά 10% στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τελευταίο ερώτημα. Ένα θέμα που δεν έχουν θέσει φυσική πόρη και η τιμή του πετρελαίου. Και τι επιπτώσεις έχει όσον αφορά τη δυνατότητα ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για την Ευρωζώνη θέσαμε το ερώτημα στον Ζαν Κλοντ Τρισέ και στον κύριο Αλμούνια, οι οποίοι μας εξέφρασαν ανησυχία, διότι η τιμή του πετρελαίου ήταν αυξημένη, ενώ η οικονομική συγκυρία ήταν κακή και ότι ήταν μεγάλος κίνδυνος αυτός που βάρινε την ανάκαμψη του 2010-2011. Θα ήθελα να ξέρω συμμεριζόστε αυτή την ανάλυση. Και τι προτάσεις έχετε για να περιοριστεί αυτός ο, ο κίνδυνος για τη μεταρρύθμιση, τη διαθεωτική οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν έχουν σαν σκοπό τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Οι μεταρρυθμίσεις που έχω υπόψη μου, κυρίως όσον αφορά την γύρανση του πληθυσμού, έχουν σαν σκοπό την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης που θα πρέπει πάση θυσία να αυξηθεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα το βάρος που προξενείται από τη γύρανση του πληθυσμού και να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την ανεργία η οποία θα αυξάνεται τους επόμενους ε, μήνες. Δεν έχω κάποια λύση γενική να προσφέρω όσον αφορά την εξέβρεση των σωστών προσεγγίσεων για να επανισορροπήσουμε τα δημοσιονομικά μας. Εκεί η σταθεροποίηση των δημοσιονομικών περνάει και από εθνικό φίλτρο. Κάθε χώρα, κάθε μέλος της Ευρωζώνης θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι καλύτεροι μέθοδοι για την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Βλέπω ότι κάποιες κυβερνήσεις τώρα αυξάνουν τη φορολογία. Βλέπω ότι άλλες χώρες μειώνουν τη φορολογία τους. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των εθνικών καταστάσεων και το πώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάθε χώρα διαφορετικά το οικονομικό πρόβλημα. Αναφέρατε δύο συγκεκριμένα μέσα, φορολογικά μέσα, κυρίως φορολόγηση των χρηματοστικών συναλλαγών. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εν ονόματι της ε, ευρωμάδας, διότι δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη θέση πάνω σε αυτό. Δεν έχω κανένα ταμπού όσον αφορά την ε, επαναφορά τέτοιου φόρου. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε να εισαγάγουμε στην Ευρώπη σε μια συγκεκριμένη χώρα τέτοιο φόρο ή αν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη τη διεθνή κοινότητα ο φόρος. Κυρίως τους ε, μεγάλους χρηματοδοτικούς κύκλους να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος. Αν θα είναι ε, φόρος τόμπιν ή κάποιο άλλο είδους φόρου. Ας συζητηθεί το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, Ευρωμάδα αυτό το θέμα. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα μέσα πώς θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και, και πώς μπορούμε να καταρτήσουμε έναν κατάλογο μέτρων αντιπίνων έναντι ε, κυβερνήσεων και δικήσεων που δεν συμμορφώνονται. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Τρισέ και του κυρίου Αλμούνια, τις συμμερίζομαι. Τι επίπτωση θα έχει αύξηση τιμής του πετρελαίου σε μια ανάκαμψη που ούτως ή άλλως θα είναι πολύ μέτρια και δειλή αυτή η ανάκαμψη. Αν ξαναυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, βλέποντας την παγκόσμια οικονομική ε, κατάσταση, θα δημιουργήσει κινδύνους. Όπως κάναμε πολλές οικονομικη κατασταση θα ξεκινήσουμε καινούριο διάλογο με τις παραγωγές χώρες για να προσπαθήσουμε κάπως να διοχετεύσουμε τις συνέπειες της αυξοτιμής, της τιμής του πετρελαίου. Για να καθησυχάσουμε όσον αφορά ενδεχόμενη μελλοντική ανάκαμψη, αν βρούμε μια σχετική λύση και διοχέτευση αυτών των αυξήσεων. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Σάντσες Περσέιδο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούνκερ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη, όταν θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Ευρωζώνης, η Ευρωζώνη θα έχει μια επίσημη διάσταση πλέον, μια θεσμική δομή. Αυτό τι θα σημαίνει, ότι θα είναι δυνατόν μια συγκεκριμένη ατζέντα της Ευρωομάδας ή θα είναι μια πιο δεσμευμένη ατζέντα προς το ΕΚΟΦΗΝ. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στην ενδυνάμει ανάπτυξη ως ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό θέτει το ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μη ισόρροπων παγκόσμιων σχέσεων και με τη διαφορετική πτυχή που έχει το κάθε κράτος μέλος ε, θα ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο αυτό στη ζώνη ευρώ. Και γι' αυτό είναι σαφές για την ενδυνάμει αυτή ανάπτυξη η μεθοδολογία είναι διαφορετική. Μία που θα βασίζεται στη ζώνη ευρώ θα μπορούσε τα θέματα της ανεργίας ε, ε, και τα θέματα κοινωνικά να τα ε, θέσει σε μεγάλη κλίμακα. Δεν είναι μόνο η ανάγκη μιας διαφοροποιημένης στρατηγικής, αλλά μιας στρατηγικής κοινή που θα επιτρέπει να δρούμε με μεγαλύτερο σθένος, δρατώμενοι του οικονομικού δυναμικού, βελτιώνοντας το μέγιστο τη δυνατότητα του να δοθούν απαντήσεις από τη Ευρωζώνης. Τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά και την ε, εξυγίανση και βιωσιμότητα αηφορία του, Είναι σαφές ότι με τον ορίζοντα της υπεργύρανσης και των προβλημάτων προβλημάτων που υπάρχουν οικονομικά είναι αναγκαίο να αποφύγουμε κάθε προσπάθεια να εξέλθουμε από την κρίση να καταλήγει σε κατηγορίες ή επικρίσεις. Πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ε, συνεπής πολιτική ευρωπαϊκή και μια πιο θα το έλεγα με θετικούς προσανατολισμούς στρατηγική δραστηριοποίηση, εξετάζοντας το αν θέλουμε να έχουμε μια παρουσία στην παγκόσμια σκηνή και όσον αφορά και την φορολογία των διεθνών αγορών κεφαλαίων που είναι ένα ε, θέμα κρίσιμης σημασίας. Ευχαριστώ. Euh, Ήδη έδωσα κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Κυρίως όσον αφορά τα φορολογικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για καλύτερη διοργάνωση του φορολογικού τοπίου την ημέρα που η Ευρωομάδα θα γίνει επίσημο σχήμα του Συμβουλίου θα εξελιχθούν τα πράγματα με πιο ενθεριντικό τρόπο από ό,τι τώρα. Αυτό θα έλεγα. Συχνά σας εξήγησα ότι είμαι πρόεδρος μιας ανεπίσημης, μιας άτυπης ομάδας. Δεν μπορώ να λέω τα πάντα προς τα έξω, δεν μπορώ να αποκαλύπτω τι συζητούμε, αλλά οι ανεπίσημες συζητήσεις εντός της ομάδας είναι χρησιμότατες για τις άλλες κυβερνήσεις που ακούν ένα συνάδελφο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι η ανταλλαγή απόψεων τροφοδοτεί τον προβληματισμό όλων επί του θέματος. Τη στιγμή όμως που θα γίνει ενήλικη η Ευρωμάδα μέσω της ε, κύρωσης της ηθίκης της Αβώνας ε, θα μπορούμε προς τα έξω να είμαστε πιο επιθετικοί, τολμώ να πω, και εγώ εύχομαι γρήγορα ε, να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας γιατί κάποιες φορές ενοχλούμε που πρέπει να σιωπώ κάποιες στιγμές που ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής και πολύ ανοιχτός και να μιλήσει κάποια πράγματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας working program στην Ευρωμάδα που καταρτίζεται για μία εξάμεινη περίοδο. Ε, μόνο μεθοδολογικές αλλαγές μπορούν να γίνουν τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Νομίζω ότι όσον αφορά τις γενικές ανισορροπίες, ε, τις παγκόσμιες ανισορροπίες, ε, έδωσα απάντηση. Συμμερίζομαι την άποψή σας. Ρεμόν Τρεμόζο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γιούνκερ. Ευχαριστώ, Σάρα. Φοβούμε για το μέλλον του ευρώ. Χτες ήρθε και ο Στρισέδο και ζήτησε συγγνώμη για το ισχυρό δολάριο. Είπε ότι Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό δολάριο. Αυτή όμως δεν είναι η επιθυμία της Federal Reserve. Είδα τα τελευταία χρόνια ότι η κινέζικη οικονομική επιτυχία θα δώσει κίνητρα σε άλλες αναδυόμενες επιχειρήσεις, ε, εταιρείες συγγνώμη, να μιμηθούν το κινέζικο σύστημα ισοτιμίων. Προβλέπω ισχυρότερο ευρώ τα επόμενα χρόνια. Και κατά την άποψή μου, ένα ισχυρότερο ευρώ θα δυσκολέψει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη που χρειαζόμαστε. Πρέπει να εδράζεται επί βιομηχανικών εξαγωγών στον υπόλοιπο κόσμο. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό κύριε Γιούνκερ. Σας ευχαριστώ. Απάντηση. Δεν μ' αρέσει αυτή η συζήτηση για αδύναμο ευρώ, για δυνατό ευρώ. Έχουμε το ευρώ. Τελεία και παύλα. Δεν μου αρέσει η έκφραση απόψεων. Δεν θέλω να εκφράσω απόψεις που σχετίζονται με την ισοτιμία δημοσία. Είναι ευαίσθητο ζήτημα. Δεν θέλω να με παραθέτουν για πράγματα που έχω πει για τις ισοτιμίες. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τις ισοτιμίες και την σχετική πολιτική ισοτιμιών. Δεν μας αρέσει η πτυτικότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Λέμε όμως ότι θέλουμε ισχυρό δολάριο. Αυτό είναι το νόημα. Και τι εννοούμε. Αναφερόμαστε στις απόψεις των Αμερικανικών αρχών που εκφράζονται από καιρούς καιρών. Όταν σχολιάζουμε τις οτιμίες και λέμε ότι καλωσορίζουμε το γεγονός ότι και η Αμερικανική κυβέρνηση και το Αμερικανικό Federal Reserve επιμένουν στο ισχυρό δολάριο. Μ' αρέσει αυτό. Μας αρέσει αυτό που λένε οι Αμερικανοί ότι το ισχυρό δολάριο ωφελεί την Αμερικανική οικονομία. Προσέξτε το εξής. Δεν ακούσαμε να λέει κάτι τέτοιο όμως πρόσφατα η Αμερικανική κυβέρνηση και θα ήθελα να την ξανακούσω τις επόμενες μέρες. Και τέλος, Λίαμ Βανκόκ. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί ζητούν και επικαλούνται μια πολιτική εξόδου. Είμαστε σε πλήρη ύφεση. Οι πολιτικές εξόδου μοιάζουν με την επιδίωξη της στρατηγικής της Αβώνας, με οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές ελέγχου των δημοσιονομικών που συνοδεύουν αυτήν. Όμω αυτή η στρατηγική που θα έπρεπε να κάνει την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου και έπρεπε να έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, έκανε τελικά την Ευρώπη την περιοχή όπου είχε τη μικρότερη ανάπτυξη στον κόσμο. Το υπογραμμίσατε προηγουμένω. Η ανάπτυξη σήμερα δεν πάει καθόλου καλά. Όλοι οι κινητήρε τη ανάπτυξη έχουν χτυπήσει κόκκινο. Οι πολιτικέ σκότωσαν την κατανάλωση, τι επενδύσει, τι εξαγωγέ. Οι εξαγωγέ υποφέρουν. Και η μείωση της ανάπτυξης που αναφέρατε οφείλεται περισσότερο στην μείωση της εσωτερικής ζήτησης που ελήψη διαθετικών πολιτικών προσφοράς που εκφράσατε υποφέρει. Το πώς χρησιμοποιείται το παραγωγικό δυναμικό. Έχουμε φτάσει ιστορικά χαμηλά, 70% απορρόφηση δυναμικού παραγωγικού δυναμικού σε κάποιες χώρες. Έλλειψη ζήτησης, ύφεση, και ίσω τελικά μέσω αυτών μειωθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγική, το παραγωγικό δυναμικό. Και οι διαθετικέ αυτέ μεταρρυθμίσει, τελικά ίσω μειώσουν ακόμα περισσότερο το παραγωγικό δυναμικό και την ανάπτυξη. Αν οι επιχειρήσεις δεν παρακινηθούν να επενδύσουν για να ανταποκριθούν σε μια ζήτηση που σήμερα είναι εντελώ άτονη. Αναγνωρίστε ο ίδιο ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν οι αυτόματοι σταθεροποιητέ, Κάτι έγινε σε δύο χρόνια. Καλό αυτό με την προπτική ανάκαμψη. Σε αυτή η περιπτώση, γιατί δεν αναφερθήκατε σύμφωνο σταθερότητα που ανέφερα συνάδελφοι. Αυτό, όπω έλεγε ο Ρωμάνι πρώτη, αυτό είναι μια ανοησία. Σε περίοδο ύφεση εμποδίζει τι χώρε να χρησιμοποιήσουν του αυτόματου σταθεροποιητέ πλήρω. Και σε περίοδο πλήρη απασχόληση δεν δίνονται κίνητρα στι χώρε να χρησιμοποιήσουν κάποια φορολογικά μέτρα για τη χρέωση. Γιατί χρησιμοποιείται αντικυκλικά μακροοικονομικά μέτρα. Δηλαδή τι λέει, όταν υπάρχει πλήρης παραγωγή, πλήρης απασχόληση, όταν χρησιμοποιείται πλήρως το παραγωγικό δυναμικό, να μην προτείνεται μια ισορροπία δημοσιονομική. Και γιατί σε περίοδο ύφεση, απ' την άλλη, να μην επιτρέπεται τη αυτή περιπτώση στι διάφορε χώρε μέλη να ε, αφήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα να λειτουργήσει για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα ανάκαμψης. Απάντηση. Καταρχάς, ποτέ δεν θεωρούσα ότι δεν θα υπήρχε ότι εάν ε, με θεωρείτε έναν από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσφοράς είναι πολύ κατά προσέγγιση η περιγραφή σας ε, πάντοτε έλεγα ότι δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο στην ε, προσφορά αλλά στην προσφορά και στη ζήτηση σχετικά με την κατάσταση την οποία έχετε περιγράψει το, το σύμφωνο σταθερότητος πρέπει να αξιολογείται για το ότι είναι. Όταν είχε πει ο κύριος Πρόντι ότι ελπάκτο το στούπιντο, νομίζω ότι ε, έτσι ήταν η συνθήκη. Το Μάρτιο του 2005 το αναθεωρήσαμε λέγοντας αυτά τα οποία εσείς ε, εύχεστε. Να υπάρχει δηλαδή ε, μία φάση προληπτική και μία φάση ε, διορθωτική. Όταν δηλαδή πάει καλά η οικονομία, οι συνθήκες μας υποχρεώνουν να μειώσουμε τις τις τις διορθωτικές παρεμβάσεις στον προπολογισμό ενώ όταν πάμε καλά μπορεί η συμφωνία να επιτρέψει να υπερβούμε το 3% πράγμα το οποίο πριν από το 2005 δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά τώρα μετά την αναθεώρηση του 2005 μπορούμε να το πράξουμε και ως εκ τούτου η επιθυμία σας έχει εκπληρωθεί πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα ελλείμματα και να ε, επιβαρύνουμε το χρέος το οποίο θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές αλλά η συμφωνία αυτή επιτρέπει κάπως το σύμφωνο ε, επιτρέπει να διευκολύνουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που παραστήκατε. Ευχαριστώ πολύ ε, για τις απαντήσεις που μας δώσατε και προτού φύγουν όλοι σχετικά με ε, την μετάφραση και τις τροπολογίες προηγουμένες εάν ε, η προθεσμία λήξης στις 8 Οκτωβρίου θα μπορέσουμε να έχουμε την ε, ανταλλαγή απόψεων στις 19 Οκτωβρίου πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είσαστε 9 η ώρα το πρωί στο Στρασβούργο την εβδομάδα του Στρασβούργου αλλά θα μπορέσουμε επίσης να συζητήσουμε και ε, για την γενική απαλλαγή ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία που ενδιαφέρει την Επιτροπή ΙΜΚΟ.